Bonjour à nouveau euh, à tous. Euh, euh, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos intervenants. Καλώς ορίσατε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Πίρσορ Οντοναχιού στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Connect στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Σαμπινσκή. Υπεύθυνο για την κοινωνική ασφάλεια στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνονται τακτικά ανταλλαγές απόψεων σε ό,τι αφορά το θέμα του του διαστήματος και το ασφάλεια για να δούμε τι ισχύει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όλοι υπόψη μας ποιες είναι οι οικονομικές ευκαιρίες που εμπλέκονται εδώ. Και η μετάβαση στο δίκτυο 5G θα αποτελέσει ε, μια ευκαιρία η οποία θα αλλάξει κατά εκβάθρον τον τρόπο λειτουργίας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε απόλυτα ενημεροί για τους κινδυνούς και τις ευκαιρίες που ε, ενέχει αυτή η καινούργια τεχνολογία. Το 5G δεν αποτελεί μόνο μια βελτίωση τεχνολογική, πρόκειται για ένα διαφορετικού τύπου τεχνολογικό τρόπο που θα επιτρέψει εντελώς διαφορετικές χρήσεις και εφαρμογές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά την εξωτερική άμυνα. Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα. Εδώ και μήνες ακούμε και παρακολουθούμε τις ε, αμερικανικές αρχές να μιλούν για το κίνδυνο απώλειας της ε, τεχνολογικής κυριαρχίας σε ό,τι αφορά και τη χρήση τεχνολογίας ε, κινηστικής προέλευσης για την τεχνολογία 5G. Εκφράζουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας ε, για τις εξέλιξεις αυτές. Γι' αυτό λοιπόν και επιλέξαμε το σημερινό θέμα για τη σημερινή ακρόαση. Κυρία Αντωναχιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξέφρασε τις ε, ανησυχίες της και την παρακολούθηση των αποδόσεων αυτών σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια. Θα υπάρξουν εθνικά μέτρα σε ένα ε, πλαίσιο αναρμονισμένο για την αξιολόγηση και στην ε, ακρόαση του ο Επιτροπός κ. ήδη μίλησε και για τους 6G υπογραμμίζοντα ότι θα επικεντρωθούμε σε τρει πυλώνε: την προστασία, την ε, μεταμορφώση και την πρόβλεψη για το μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να μπορείτε να μα επισημάνετε πω ε, σκοπεύουμε να κατακτήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε ό,τι αφορά το 5G. Ο Σωτήγος Σαντίνσκι θα θέλαμε να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής για το πώς έχουν ε, τα πράγματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, να δούμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι μηχανισμοί συντονισμού προκειμένου να εφαρμοστούν μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχά στον κύριο Ντοναχίου. Merci, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Euh, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ που μα επιτρέπετε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό θέμα θα υποθέσω ότι κάποια πράγματα τα γνωρίζετε, αν δεν τα γνωρίζετε διορθώστε με. Η λειτουργία του δικτύου 5G στην Ευρώπη ήταν στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση λόγω της σημασίας που έχει για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό ήταν η βάση του προγράμματος δράσης 5G που ξεκινήσαμε το 2016. Να δώσουμε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη του 5G με στόχο να έχουμε μία ταυτόχρονη ανάπτυξη υπηρεσιών 5G σε όλα τα κράτη-μέλη, ξεκινώντας από φέτος και πλήρη ε, λειτουργία το 2025. Φιλόδοξο στόχο. Το πρόγραμμα δράση στηρίζεται στο ότι τα 5G αλλάζει το παιχνίδι. Δεν είναι μια ταχύτερη εκδοχή των 4G, αλλά είναι μια νέα προσέγγιση πλατφόρμας που εξασφαλίζει όχι μόνο ταχύτερες τεχνολογίες, αλλά μεγαλύτερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων και αξιοπιστία και του σήματος και της μεταφοράς των δεδομένων και του χρόνου αντίδραση σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η βάση των γνώσεων για το 5G. Έχει επιπτώσει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όχι μόνο την τεχνολογία και την πληροφορική, γεωργία, μεταφορές, ενέργεια, μέσα ενημέρωσης, ψυχαγωγία κτλ. επηρεάζονται. Θα επηρεάσει την λειτουργία Τη ε, της ρομποτικής, της λειτουργίας των εργοστασίων, την διαπίστωση σφαλμάτων στα δίκτυα ενέργειας κλπ. Λόγω ακριβώς του ρόλου του, ε, των 5G υπάρχει μια αυξανόμενη επίγνωση της στρατηγικής ευαισθησίας που αντιπροσωπεύει αυτή η τεχνολογία για την οικονομία και την κοινωνία. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και ενισχύεται μια συζήτηση για το κίνδυνο να εξαρτώμεθα υπερβολικά για κάποια στοιχεία του δικτύου από το εξωτερικό. Και αυτό είναι το ζήτημα της ασφάλειας. Η διάσταση ασφάλειας των 5G και τα μεγάλα πλεονεκτήματα βεβαίως ε, της ε, τεχνολογίας ε, αυτής που παρέχουν τεράστια ικανότητα κρυπτογράφησης των δικτύων. Στις 3 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο υιοθέτησε τα συμπεράσματά του για τη σημασία ε, του 5G κυρίως από την οπτική της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους. Εμείς καλωσορίσαμε τα συμπεράσματα που συνδέει την κυβερνοασφάλεια με την οικονομική δύναμη του 5G, εξασφαλίζοντας ότι θα έχουμε μια σαφή εικόνα πως η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και η παροχή εξοπλισμού για πρόσβαση στο 5G είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό θα αποκτήσει και γεωπολιτική σημασία καθώς το 5G έρχεται στην κορυφή της πολιτικής ημερήσιας διάταξης. Η απάντηση για τις προκλήσεις αυτές που έγιναν ήδη πέρυσι το, Μά, το Μάρτιο ε, οδήγησε την Επιτροπή να εκδώσει μία σύσταση για την κυβερνοασφάλεια και τα 5G. Με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου πρέπει να σας πω. Το πρώτο βήμα ήταν να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να κάνουν μια δική τους εθνική αξιολόγηση κινδύνων. Αυτό έγινε με τεχνική υποστήριξη και βοήθεια της Επιτροπής της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας της ΕΝΙΖΑ. Κατόπιν, αφού συμπιλήσαμε το κείμενο, δουλέψαμε τα κράτη-μέλη για να ετοιμάσουμε το τελικό κείμενο που δημοσιεύτηκε πέρσι τον Οκτώβριο. Το επόμενο βήμα, όπω είπε η πρόεδρο, είναι η εργαλειοθήκη που ετοιμάζουμε με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ε, να τονίσω επίσης ότι η δουλειά που κάναμε στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας σημαίνει ότι ε, ασχοληθήκαμε με την τεχνική διάσταση της ασφάλειας εδώ και κάποιο καιρό. Είχαμε ε, μια, ε, δημόσια, μια ΣΔΙΤ ε, για τον τομέα αυτό στο πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο και ένα work stream σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που παρακολούθησαν την εξέλιξη αυτή στα πλαίσια της ομάδας εργασίας ασφάλειας και σε συνεργασία με συγκεκριμένα project. Ιδίως το πρόγραμμα Ensure 5G, 5G που κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου εντοπίζοντας τις περιπτώσεις που είναι ευάλωτες. Πέραν λοιπόν των εθνικών και της ευρωπαϊκής αξιολόγησης κινδύνου, ομόφωνα τα κράτη-μέλη υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεργαστούν και να ασχοληθούν σοβαρά, ουσιαστικά σοβαρά με το θέμα. Αυτό είναι η βάση της δουλειάς που κάνουμε τώρα, που αποκαλούμε εργαλειοθήκη μετριασμού του κινδύνου δηλαδή μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη-μέλη έναντι εντοπισμένων, εντοπισθέντων κινδύνων ή κινδύνων που αξιολογούνται ως σημαντικοί. Αυτό θα επιτρέψει την Ένωση να μιλήσει με ενιαίο τρόπο στα θέματα ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας. Η συνεργασία των κρατών είναι καθοριστική και εμείς θα επιτρεψει στην ενωση να μιλησει με ενιαιο τροπο στα θεματα ασφαλειας ασφαλειας αυτή τη δουλειά στην ομάδα εργασίας για την ε, οδηγία δικτύου, ασφάλειας δικτύων ένα πλαίσιο εξαιρετικά χρήσιμο. Τώρα, τι γίνεται στο μέλλον. Ποια θα είναι η χρήση, οι τομείς που θα καλυφθούν από αυτό. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη δεδομένου του στρατηγικού ρόλου που παίζουν τα 5G, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την βιομηχανική παρουσία Ευρωπαίων, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα του συστήματος, όπως, του συστήματος. όπως ξέρουμε ήδη, δύο στους τρεις μεγαλύτερους προμηθευτές ε, ε, στα δίκτυα είναι Ευρωπαίοι, είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να υποστηρίξουμε την κατάσταση αυτή. Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως δεν εξασφαλίζει επιτυχία ή ασφάλεια προμήθειας. Πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε, να παράξουμε και να εξασφαλίσουμε τις τεχνολογίες εν ώψη και τη σημερινή ε, πραγματικότητα και του μέλλοντος. Ένα βασικό θέμα που θα συζητηθεί εδώ αφορά τα θέματα πιστοποίησης και τυποποίησης. Με βάση τι κρίνουμε την ασφάλεια, τη δυνατότητα ασφάλειας ή τον κίνδυνο ασφάλειας ενός ε, ε μηχανισμού. Ήδη στο συντονισμένο, στη συντονισμένη αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνουμε μια σειρά ε, ζητημάτων ασφάλειας. Αυτό ωστόσο είναι ουσιαστικό. Δίνουμε έμφαση στο σημείο αυτό καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν όρια στα, στις δυνατότητες αυτές. Τα κράτη-μέλη λοιπόν συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα αυτό, ιδίως έχουμε, ιδίως έχουμε στα θέματα πιστοποίησης ακόμα, πώς θα γίνεται η πιστοποίηση. Συνεργαζόμαστε με τους παραγωγούς και τον κλάδο στον τομέα αυτό και με τους επιμέρους κλάδους ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που έχουν και σημαντικούς κινδύνους αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αντιμέτρων. Προσπαθώντας να παράσχουμε ένα σημείο αναφοράς για την πιστοποίηση ιδίως, την τυποποίηση συγγνώμη, ιδίως των υπηρεσιών ε, κυβερνοασφάλειας. Θα ήθελα να να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ζήτω συγγνώμη προς όλους. Ιρλανδός είμαι, ξέρετε, και έχω προβλήματα όταν μιλάω στα αγγλικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς μιλάω πολύ γρήγορα γιατί φοβάμαι τα αγγλικά μου. Η Επιτροπή εμπλέκεται προφανώς στο παγκόσμιο πλαίσιο τυποποίησης. Για να σας μπερδέψω ακόμη περισσότερο, η τυποποίηση γίνεται στα πλαίσια μιας ομάδας που λέγεται 3GPP, δηλαδή ομάδας τυποποίησης των 3G, αλλά γιατί ξεκίνησε την εποχή που είχαμε τα 3G. Υποστηρίζει τους εμπλεκόμενους φορείς, μετέχει η ίδια. Αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που σημαίνει ότι η Ευρώπη παίζει ένα συνεχιζόμενο ρόλο σημαντικό και σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση αυτή. Τώρα έχουμε ξεκινήσει να συζητούμε και το θέμα των 6G, του, της, της έκτης γενιάς. Καθώς λοιπόν αρχίζουν και έρχονται τα αποτελέσματα από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο από το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και από την υλοποίηση του δικτύου πέμπτης γενιάς, θα συμμετέχουμε ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να αγνοούμε ότι πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με τις επόμενες γενιές. Θα μου πει κάποιος ακόμα δεν ξεκινήσαμε την πέμπτη γενιά θα συζητάμε την έκτη. Αυτό όμως είναι σημαντικό για να, το, για να μπορέσει η Ευρώπη να είναι πάντα στην πρωτοπορία. Η πέμπτη γενιά εντάσσει και ενσωματώνει μια σειρά νέων λειτουργιών. Η έκτη γενιά μπορεί να λάβει υπόψη άλλες παραμέτρους, το ίντερνετ των πραγμάτων και ελπίζουμε ότι καθώς πηγαίνουμε προς την έκτη αυτή γενιά θα υπάρξει μια ενοποιημένη αδιάλειπτη πλατφόρμα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο που θα παρακολουθείτε ταυτόχρονα από ε, υπηρεσίες καταστολής, από υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και από την ασφάλεια του δικτύου, ούτω ώστε να παράσχει και ασφάλεια στο δίκτυο και ασφάλεια στα άτομα. Αυτή είναι η φιλοδοξία που εκφράσαμε. Στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείνουμε μία νέα θεσμική εταιρική σχέση, Smart Networks and Services λέγεται, που θα ασχολείται με την έκτη γενεά, το 6G. Εμείς με το Κοινοβούλιο λοιπόν συνεργαζόμαστε για να αρχίσει να λειτουργεί με ασφαλή τρόπο το δίκτυο πέμπτης γενιάς. Παράλληλα κάνουμε πολλή δουλειά και στην έκτη γενιά. Αυτή είναι η ουσία της νέας μας στρατηγικής σε ό,τι αφορά αυτές τις νέες τεχνολογίες. Να μιλήσω λίγο τώρα για το θέμα που θέσατε, την ασφάλεια. Δεν είμαι ειδικό, ούτε μπορώ να μιλήσω για τον ε, ειδικό ρόλο της 5ης γενιάς στα θέματα άμυνας. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ε, παράμετροι άμυνας στο 5G, εμείς δουλεύουμε κυρίως στα στο μη στρατιωτικό ρόλο του 5G, αλλά ξέρω ότι θα έχω, και μπορώ να σας πω από αυτήν την οπτική, ότι θα έχει τεράστια επίπτωση στην λειτουργία των δορυφόρων. Θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την ευρυγονική υψηλής ταχύτητας κάλυψη όλης της Ευρώπης. Είμαι βέβαιος ταυτόχρονα ότι πολλές παράμετροι του 5G που σχετίζονται με τις υποδομές, τις μεταφορές κλπ. θα γίνουν ασφαλέστερες όταν εισαχθεί η δορυφορική συνιστόσα του 5G και του μετά τα 5G. η ποσοτικοποιημένη αυτή ανάπτυξη θα έχει θετικές συνέπειες στην ασφάλεια. Βέβαια, έχω πολλούς συναδέλφους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα και μπορούσαν να σας ενημερώσουν για αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω κλείνοντας ότι η Επιτροπή κυρία Βαντελάιν υπογράμμισε το ρόλο των, της πέμπτης γενεάς, ιδίως των προτύπων για την τεχνολογία πέμπτης γενεάς δουλεύουμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε να παράσχουμε ως Νέα Επιτροπή ένα σύνολο πολιτικών που θα καλύψουν τον τεθέντα στόχο και θα παράσχει ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια στο τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο στρατηγός κ. Σαμπίνσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο και να τοποθετηθώ για τις προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας και άμυνας που θέτει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς ή το δίκτυο δεδομένων πέμπτης γενιάς με δεδομένο ότι το περιβάλλον ασφαλείας είναι πολύ περίπλοκο, πολύ απαιτητικό και αλλάζει συνεχώς, θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική με μια πιο κοινή, πιο αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων CSDP. Ε, πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να έχουμε τεχνολογία και συστήματα για την επικοινωνία και την πληροφορική που θα αγγιώνται την διαθεσιμότητα και την ακαιρεότητα των δεδομένων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλες οι δυνατότητες εξαρτώνται από το εμπιστευτικό, από το απόρριτο, από την ακαιρεότητα και από τη διαθεσιμότητα αυτών των συστημάτων. Είναι προφανές σε όλους μας ότι οι στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις CSDP ασφάλειας και άμυνας εξαρτώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ευέλικτες υποδομές και υπηρεσίες στο θέμα αυτό, οι οποίες όμως να μπορούν να προστατευτούν και να μπορούν να ε, είναι αποτελεσματικές. Μπορούν έτσι οι στρατιωτικοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που τους έχουν επιφορτήσει οι πολιτικοί ηγέτες. Το στρατιωτικό επιτελείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, ο βασικός εταίρος για τέτοιου είδους δραστηριότητες και είναι ουσιαστικά ο στρατιωτικός ε, πελάτης και πρέπει να διασφαλίσει και την κυβερνοασφάλεια και πρέπει να σχεδιάσει, να καθοδηγήσει και να παρακολουθήσει του σύνεγγυ στην εφαρμογή όλων αυτών των δράσεων ε, και των λύσεων για να έχουμε κυβερνοάμυνα και κυβερνοασφάλεια πρέπει να προσδιορίσουμε τις στρατιωτικές απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις για τις σχετικές αποστολές και επιχειρήσεις και να στηρίξουμε ε, το στρατιωτικό δυναμικό και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των λύσεων. Τα μέτρα ε, πρέπει να είναι τα κατάλληλα. Άρα πρέπει να διενεργηθεί η μελέτη αξιολόγηση κινδύνου και να υπάρξει η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όπου χρειάζεται. Οφείλω να τονίσω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τεχνολογικές συστάσεις, ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε τις πολιτικές και οικονομικές πτυχές της πέμπτης γενιάς, των δικτύων πέμπτης γενιάς, του 5G. Μπορούμε όμως να παρέχουμε τις βέλτιστες δυνατές στρατιωτικές συμβούλες. Έχουμε νέες τεχνολογίες ανατρεπτικές, και στα στρατιωτικά αλλάζουν το περιβάλλον εργασία μας και μάλιστα με ταχύς ρυθμούς και ε, σε εναρείο επίπεδο και σε χερσαίο και σε θαλάσσιο επίπεδο ε, λειτουργούμε ε, και τα καθοδηγούμε όλα αυτά με ηλεκτρονικό τρόπο, με πολύ περίπλοκες υποδομές. Ακόμα και το πεζικό το καθοδηγούμε με πολύ περίπλοκες ηλεκτρονικές υποδομές και μοιραζόμαστε τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα σε πραγματικό χρόνο. Όλο και περισσότερο βασιζόμαστε σε τέτοιου είδους λύσεις οι οποίες διατίθενται στην αγορά, εμπορικές λύσεις για να λειτουργήσουμε στρατιωτικά. Άρα ε, όλη αυτή η ψηφιοποίηση ε, του πεδίου μάχης και της ε, συνδεσιμότητας είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας. Και θα εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνολογία 5G. Αυτό είναι προφανές. Δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την εξάρτησή μας από την πέμπτη γενιά γιατί χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της πληροφορικής, της επικοινωνίας των πληροφοριών και για στρατιωτικούς σκοπούς. Και οι φορείς και οι πάροχοι είναι μη στρατιωτικοί και προσπαθούν να στηρίξουν και τη στρατιωτική κινητικότητα οι στρατιωτικές υπηρεσίες ε, πληροφορικής συνδέονται με ε, ε, εμπορικούς παρόχους που δεν είναι στρατιωτικοί, ανήκουν στο, στους, στις πολιτικές οντότητες. Για παράδειγμα, όσοι χειρίζονται τους δορυφόρους. Οι δορυφόροι, βασιζόμαστε στους δορυφόρους για τα στρατιωτικά, αλλά τον δορυφόρο το λειτουργεί εμπορικός πάροχος και όχι στρατιωτικός. Δημιουργούνται λοιπόν δε ζητήματα κυβερνοασφάλειας ε, πολύ πιο περίπλοκα πέρα από τα ίδια υφιστάμενα και πρέπει να μετριάσουμε αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα στρατιωτικά μας καθήκοντα. Απάξω όμως και ε, τροποποιηθεί και προσαρμοστεί η τεχνολογία 5G για στρατιωτικούς σκοπούς για να μπορεί να τη στηρίξει, να στηρίξει τις στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Ε, ο ίδιος ο στρατός είναι, έχει λίγες ευκαιρίες να διαχειριστεί τέτοιου είδους λύσεις για να εγγυηθεί την ασφαλή χρήση αυτής της τεχνολογίας. Επομένως, αυτά τα μέτρα μετριασμού, οι διατάξεις μετριασμού των επιπτώσεων πρέπει να είναι οικονομικού, πολιτικού χαρακτήρα ή βιομηχανικού. Δηλαδή, αξιολογώντας το 5G πρέπει να καταλάβουμε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκφύσεως λόγω της ιδιαιτερότητάς τους σε θέματα ε, εμπιστευτικότητας, απορρίτου, ακαιρεότητας ε, των συστημάτων ελέγχου και διοίκησης απαιτούν λοιπόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις υψηλότερο επίπεδο κυβερνοασφάλειας και μια κυβερνοεπίθεση σε στρατιωτική βασικές ηλεκτρονικές ε, υποδομές ε, μέσα από το 5G θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλες τις επιχειρήσεις και να οδηγήσει και σε απώλεια ανθρωπίνων ε, ζωών αυτό το ενδεχόμενο. Άρα μπορεί να μην μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, να αποτύχουμε δηλαδή και αυτό θα έχει πολύ σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Άρα πρέπει να έχουμε μέτρα αντιμετώπισης συνολικά, περιεκτικά και με βάση τα κοινά πρότυπα για την ασφάλεια θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέξει τους παρόχους 4G και 5G. Οι πάροχοι θα πρέπει να κληθούν να αποδείξουν την πλήρη τους ανεξαρτησία από, μη, ε, ε, από κυβερνήσεις και παράγοντες άλλους που δεν ε, εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός ΕΕ. Ακόμα και αν αποδειχθεί αυτό και αν, ακόμα και αν ο στρατός αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στο 5G, Δηλαδή, λόγω σχεδιασμού, χάρη στο σχεδιασμό να καταστεί η τεχνολογία 5G ασφαλής, η διαχείριση του δικτύου θα γίνει πολύ πιο περιπλοκή για μας. Γιατί όντως θα αυξήσει τον αριθμό των εταίρων, των εμπλεκόμενων μερών που συμμετέχουν. Οι παρόχοι υλικού και λογισμικού θα έχουν πιο κεντρικό ρόλο να διαδραματίσουν και θα μεταβιβάζεται ο έλεγχος δικτύου σε, μια, σε εταιρείες και σε λύσεις που διαχειρίζονται το λογισμικό αυτό αυτό. και αυτό από μόνο του ως γεγονός αποτελεί πρόβλημα κυβερνοασφάλειας. Ήδη ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πρόκληση για την άμυνα. Εάν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων και βάλουμε και άλλους στο παιχνίδι, αναγκαστικά λόγω του 5G, ε, θα είναι πολύ πιο δύσκολη η δουλειά μας. Και τέλος περιμένουμε να είναι πολύ περίπλοκη αυτή η κατάσταση και αυτή η περιπλοκότητα θα βαίνει αυξανόμενη και άρα θα χρειάζεται όλο και πιο ε, προσωπικό, αν θέλετε, με ειδικέ δεξιότητες και καταρτήσεις για να μπορέσει να τα παρακολουθεί όλα αυτά αυξάνονται δηλαδή οι δυσκολίε σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, δυσκολίε που αντιμετωπίζει ήδη οποιαδήποτε αμυντική οργάνωση στρατιωτική σήμερα. Συμπερασματικά, η τεχνολογία 5G και η ενδυνάμει χρήση της σε ε, ε, στρατιωτικές αποστολές ε, και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ε, είναι τεχνολογίες αυτές οι οποίες ε, συνοδεύονται από διάφορες προκλήσεις που θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Σβέν, παρακαλώ, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, κύριε, κυρία Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα να απευθύνω στον κύριο Ντόναχιου. Ορισμένες φορές ε, θίξατε ε, την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε ό,τι έχει να κάνει το 5G. Μιλούμε για τη στρατηγική αυτονομία και την ευρωπαϊκή ε, κυριαρχία σε ό,τι έχει πολύ συχνά. Τι εννοείτε εσείς, εννοείτε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόνομα να μπορεί να δράσει χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε κρίσιμους παρόχους που, παρέχουν, που βρίσκονται στις Πολιτείες ή που προέρχονται από αυτές. Να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα δηλαδή και τεχνολογικά σε επίπεδο υποδομών. Αναφέρεστε και στην Κίνα. Θέλουμε να έχουμε κυριαρχία πλήρους κλίμακας ανεξαρτητός του τι κάνουν οι Αμερικανοί σε αυτό το τομέα. Σίγουρα η τεχνολογική ηγεμονία η κινέζικη δεν θα ήταν καλό ενδεχόμενο για την Ευρώπη αν και εφόσον συμβεί. Δεν θα ήταν αυτό ε, καλό. Δεν θα μας επέτρεπε να λειτουργούμε ασφαλή συστήματα πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, οι Κινέζοι θέλουν να είναι, ηγετικοί, να είναι ηγέτες, να έχουν ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών 5G και βασίζονται σε άλλα μέρη, σε τρίτα μέρη για να τους παρέχουν τις ορισμένες συνιστώσεις αυτού του πλέγματος του 5G και οι Αμερικανοί έχουν συστήματα Android λειτουργικά από την άλλη τι επιδιώκουν, θέλουν οι ίδιοι να είναι κυρίαρχοι και απολύτως ανεξάρτητοι και αυτόνομοι, να πρέπει να, να, να μην χρειάζεται να βασίζονται του Ευρωπαίου Ευρωπαίους, ούτε στου ε, Αμερικανούς, ούτε στους Νοτιοκορεάτες, ούτε σε κανέναν άλλο εμπλεκόμενο μέρος για την παροχή κάποιου τμήματο αυτή τη αλυσίδα για το 5G. Ή μόνο το 5G αυτό καθεαυτό θα πρέπει να μας απασχολεί και όχι τα, τα υπόλοιπα τα της τεχνολογίας. Ευχαριστώ, θα ακούσουμε και τους άλλους βουλευτές και θα απαντήσετε ε, στη συνέχεια σε όλους ομαδικά. Ο Κρίς Πέτερς για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για αυτή την ενημέρωση που μας έκαναν για το 5G, για την πέμπτη γενιά. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι το 5G έχει πολύ μεγάλο οικονομικό δυναμικό, έχει περικλεί πολλές δυνατότητες σε επίπεδο οικονομίας, αλλά αποτελεί και πρόβλημα ασφάλειας, αποτελεί και πρόκληση για την άμυνα. Είναι θέμα αυτό και στο ΝΑΤΟ και στη Europol έχει τεθεί. Και δηλαδή για τις αστυνομικές αρχές ε, της κάθε χώρας που προσπαθούν να καταδιώξουν τους εγκληματίες. Ε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφαλείας με το 5G λοιπόν σε αυτή την άσκηση. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα της άμυνας, της εθνικής ή της ευρωπαϊκής. Βέβαια σίγουρα το 5G έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια και μπορώ να σας πω ότι στο Βέλγιο πρόσφατα ε, παρακολουθήσαμε ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα, πολύ εύγλωτο. Μια πολύ γνωστή εταιρεία, η Pick and All, ε, έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης ε, και αυτό είχε πάρα πολλές συνέπειες αρνητικές. Ήταν, ε, απασχόλησε πρόσφατα τη βελγική επικαιρότητα, θα το έχετε ακούσει το θέμα αυτό. Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι όντως η κυβερνοασφάλεια είναι εθνική αρμοδιότητα, το είπατε κι εσείς. Και σήμερα πλέον αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινάει η συζήτηση για την κυβερνοασφάλεια, για την πιστοποίηση των παρόχων, τα κράτη-μέλη όμως αποφασίζουν, το καθένα. Και αυτό το ζήτημα δεν είναι πρόβλημα μόνο όταν συζητούμε την κυβερνοασφάλεια, αλλά είναι και πρόβλημα όταν μιλούμε για γεωπολιτικά ζητήματα. Και ο συνάδελφο από του σοσιαλιστέ έθιξε ε, το θέμα τη Κίνα, τη Νότια Κορέα και το καθεξή. Δεν είναι δηλαδή μόνο τεχνική η συζήτηση. Η συζήτηση για την κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο τεχνική για την ασφάλεια αυτή αυτή, είναι και πολιτική για, τις, για τα γεωπολιτικά ζητήματα που μας απασχολούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και οφείλω να πω ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικά της Ευρώπης να λέει ότι εντάξει κάποια πράγματα θα τα κάνουμε, κάποια θα τα βάλουμε, ε, θα περιλάβουμε, θα θεσπίσουμε επιστοποιήσεις και το καθεξής, αλλά μέχρι εκεί και τα υπόλοιπα τα σοβαρά θα τα κάνουν τα κράτη-μέλη γιατί υπάρχει εθνική αρμοδιότητα αρμοδιότητα και κυριαρχία, ε, τότε το πρόβλημα της ασφάλειας παραμένει εξίσου φλέγων και επίγον. Άρα τίθεται το ερώτημα, ε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ότι τώρα. Εγώ νομίζω ναι και πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί, να λειτουργήσουμε και να σκεφτούμε πιο δημιουργικά. Πρέπει να εγγυηθούμε τους κανόνες για την αγορά, τις διεθνείς αγορές, να αποφύγουμε τα μονοπόλια και να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει παραβίαση ε, και παράβαση μάλλον των κανόνων για τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ίσως το ζήτημα της ασφάλειας, της ασφάλειας και το, του 5G να μπορούμε να το χειριστούμε με τα υφιστάμενα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, έχω την εντύπωση και αυτό ρωτώ να μου επιβεβαιώσετε ότι προς το παρόν δεν έχουμε βρει σωστές απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λύσουμε οριστικά το θέμα ασφαλείας και άμυνας και να απαντήσουμε στα ερωτήματα του ΝΑΤΟ από τη μία και δεν έχουμε λύσει και το πρόβλημα της ασφάλειας σε σχέση με την αμυγή αγκληματικότητα που απασχολεί τις αστυνομικές αρχές και τη Europol. Ευχαριστώ κύριος Μπασέσκου. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Είναι σαφές ότι το 5G θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ μεγάλη βελτίωση της οικονομίας. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι αναφορικά με τα νέα κράτη-μέλη να καλύψουν την ε, απόσταση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σε σχέση με τα παλιά κράτη-μέλη. Το σύστημα λοιπόν αυτό θα δώσει ευκαιρίες για ταχύτερη ανάπτυξη. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγγυηθεί μία λύση για να υπάρξει ίση κατανομή του 5G σε όλα τα κράτη-μέλη. Εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα. Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες διερωτώνται και χρειαζόμαστε μία απάντηση από αυτού. Θα δημιουργηθούν προγράμματα για ίσες ευκαιρίες σε όλα τα κρατη Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέτσος. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Και φαίνεται ότι χάσαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στον αγώνα του 5G. Αλλά προετοιμαζόμαστε για να συμμετέχουμε στον αγώνα για το 6G. Την έκτη γενιά. Διαβάζοντας όμως τον διεθνή τύπο, φαίνεται ότι οι Κινέζοι έχουν επενδύσει πάνω από 60 ευρώ, ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά κερδολογικές πιστώσεις, κρατικές επιδοτήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν το σύστημα 5G. Ωραία λοιπόν, θέλουμε να περάσουμε στο συστημα 6 έκτης γενιάς, 6G. Πόσο θα κοστίσει όμως αυτό. Θα υπάρξει διαθεσμική συμφωνία, συνεργασία. Το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι συζητάμε ωραία και καλά, χωρίς όμως να χρηματοδοτούμε τελικά τίποτα. Ο κ. Αντώνοχιου θα μπορούσε να μας δώσει πιο πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοοικονομικές προπτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Εφόσον, με δεδομένου ότι η Κίνα έχει δαπανά τεράστια κονδύλια για την ενίσχυση του 5G, ενώ εμείς ε, θέτουμε κάποια ζητήματα αγοράς ενώπιον μιας τεράστιας προκλήσεως ε, όπου χρειαζόμαστε το αντίθετο, ένα όραμα, ένα μεγάλο όραμα και μια ουσιαστική στρατηγική αυτονομία, μια ευρωπαϊκή κυριαρχία στην πράξη στο μέτωπο αυτό. Εμείς ποτέ δεν προτείναμε στον ΠΟΕ να αναθεωρήσει τους κανόνες της αγοράς αυτής με βάση το δεδομένο ότι είναι τόσο ανισόρροπη η σχέση η, εν, ε- της, Ένωσης και των κρατών μελών σε σχέση με την Κίνα. Αν ισχύει αυτό, ε, η πέμπτη γενεά είναι ένας από τους πολλούς τομείς όπου η δυνατότητα απόκτησης ε, ευρεσιτοχνιών σε, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο σκιάζει το μακροχρόνιο όφελος για την κοινωνία. Για αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία ουσιαστική εμπλοκή μας στο χώρο των 5G και της διπλής χρήσεώς του για να προστατευτούμε καλύτερα από μία πιθανή επίθεση. Κάνουμε αυτό που χρειάζεται ή χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει και θα βοηθά τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν την αυτονομία λήψη απόφαση στον τομέα αυτό. Χρειαζόμαστε ένα εθνικό πλαίσιο και ένα ευρωπαϊκό επιστέγασμα. Τελευταία ερώτηση. Είναι πραγματικό ότι οι Κινέζοι είναι τόσο μπροστά στην τεχνολογία. Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι πιο μπροστά από τους Κινέζους και πρέπει να τους υποστηρίξουμε και να τους προβάλλουμε. Ευχαριστώ κυρία Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου, κυρία Φωτιγκά. Υπάρχουν πολλοί μύθοι για το θέμα αυτό. Και προφανώς ε, το 5G σημαίνει τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης τεχνολογικής εξέλιξης αλλά προφανώς και συνεπάγεται και μεγάλες προκλήσεις. Είμαστε στην ε, Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και προφανώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην πτυχή της ασφάλειας σε ό,τι αφορά το 5G και στον τομέα πρωταρχικής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ε, ασφάλειας και της άμυνας. Αναφέραμε την κυβερνοασφάλεια ως τον πρώτο και βασικό τομέα συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανώσεων. Και ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάσουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί με τη συνεργασία των δύο οργανώσεων και στην ε, διακήρυξη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και στην σχετική ε, δήλωση που έγινε. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε λοιπόν όλα τα θέματα, όλα τα ζητήματα στη μερίσια διάταξη και προφανώς ε, πολλές χώρες παρακολουθούν τις εξέλιξεις στην Κίνα και ανησυχούν. Και αυτό σαφώς και θα πρέπει να αποτελέσει ένα θέμα προς εξέταση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν τίθεται μόνο το θέμα της ε, ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά την πολιτική χρήση των εφαρμογών αυτών. Υπάρχει και μια τεράστια διάσταση ως προς την ασφάλεια, λαμβάνοντα υπόψη και την ανάπτυξη δυναμικού στρατιωτικού από πλευρά τη Κίνα. Ευχαριστώ, ο κύριος Μπούκνερ. Και θα κλείσει το σημείο αυτό ο κατάλογος των ομιλητών για τις ερωτήσεις, για να έχουμε χρόνο και για τι απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη προηγουμένω αναφερθήκαμε εν συντομία στο γεγονό ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι τόσο πολύ ε, σε ό,τι αφορά τις παράνομες ε, μεταφορές δεδομένων, αλλά και με τις νόμιμες μεταφορές δεδομένων. Να έχετε υπόψη σας ότι στον πολιτικό κλάδο, όχι στο στρατιωτικό κλάδο, υπάρχουν ε, πολλές εταιρείες που ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών θέτουν ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Η Google, για παράδειγμα. Αυτό πληττεί και τον στρατιωτικό κλάδο εν μέρη, αλλά θα ήθελα να αναφέρω την Cambridge Analytica για να σας πω πόσο ε, σημαντικό είναι το πρόβλημα που έχουν, ε, θα έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα των ατόμων με την τεχνολογία 5G. Και παρόλα αυτά, η Cambridge Analytica έχει επηρεάσει με αυτή την πρωτόγονη, αν θέλετε, μεταφορά δεδομένων ήδη τόσα πολλά άτομα. Έχουν ε, πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία όχι μόνο οδηγούν σε παρακολούθηση των πολιτών αλλά και σε πλήρη έλεγχο αυτών. Και εδώ τίθεται το θέμα και του στρατιωτικού κλάδου, τον τομέα των μυστικών υπηρεσιών, τεχνολογίες παρακολούθησης, όλα αυτά προφανώς και παίζουν ένα ρόλο. Και αυτό που θέλω να πω στη τελική ανάλυση είναι το εξή ότι θα πρέπει κατεπηγόντως να υπάρξει ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταρτιστεί τέτοια νομοθεσία γιατί οι Αμερικανοί φίλοι μας προφανώς και θα αντιταχθούν σε τέτοια ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά δεν θα το αποφύγουμε θεωρώ και για στρατιωτική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Σουντόναχιου. Να είστε καλά. Οι ομιλίες οι ερωτήσεις σας δείχνουν πόσο καλά γνωρίζετε και το πολιτικό και το τεχνικό στοιχείο. Αυτό για το οποίο εκλεγήκατε άλλωστε. Σε κάποιες ερωτήσεις θα δώσω πιο τεχνοκρατική απάντηση. Κάποια πράγματα είναι σαφή ωστόσο. Πρώτον, η σύσταση της Επιτροπής δεν είχε στόχο συγκεκριμένη χώρα ή επιχείρηση. Καλύπτει όλες τις χώρες, όλες τις επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει την ακαιρεότητα του δικτύου 5G. Δεν είχαμε στόχο να αποφύγουμε να δακτυλοδεικνύουμε κάποιους το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι η ασφάλεια απαιτεί να καλύπτονται όλοι οι εμπλεκόμενοι. Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και παντού. Όπως η Επιτροπή τόνισε σαφώς, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ανοιχτή. Είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε στην εσωτερική μας αγορά όποιον θέλει, ο οποίος όμως όχι μόνο θα σέβεται τους κανόνες, θα φαίνεται ότι σέβεται τους κανόνες και θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που ζητούμε για την ασφάλεια του δικτύου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Βεβαίως θα, ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Τα κράτη-μέλη μας λένε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αν μας πούν ότι υπάρχουν κίνδυνοι πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό έχουμε την εργαλειοθήκη που αφορά επίσης όλα τα κρατημέλη. Αυτό ήταν το προφίλ κινδύνου που θέλαμε. Κάθε πιθανό κίνδυνο. Η... η νομοθεσία για την κυβερνοασφάλεια είναι κάτι που έρχεται από μια μακρά περίοδο ενασχόλησής μας με το τομέα αυτό. Αυτό που τονίζουμε εδώ είναι ή συγκεκριμένοι κρατικοί φορείς. Η σχέση δηλαδή συγκεκριμένων επιχειρήσεων με την κυβέρνησή τους ή τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας ή πληροφοριών των συγκεκριμένων χωρών και κατά πόσον ο εξοπλισμός ε, τηρεί τα υψηλά πρότυπα. Αυτά που είπε ο στρατηγός ότι τώρα σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή βάση 40 δίκτυα γίνονται update κάτι που δίνει στον πάροχο των προϊόντων αυτών μία μόνιμη, ένα μόνιμο τελείως ε, ιδιαίτερο και, ε, και έντονο ρόλο. Άρα καθιστά τον πάροχο ε, δυνάμει θύμα τέτοιων κυβερνών ε, Για το λόγο αυτό, ο ρόλος του κρατικού φορέα που μπορεί να έχει πάρει οδηγίες από μια κυβέρνηση να ασκήσει κάτι που είναι παράνομο πρέπει να υφίσταται κυβέρνο ε, ε, αξιολόγηση κυβέρνο ασφάλειας. Η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους βέβαια. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν συνεργαστεί από κοινού χωρίς πρόβλημα και ζήτησαν από την Κομισιόν να παίξει ένα ρόλο επιπλέον και αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πάμε η κυβερνοασφάλεια δεν είναι θέμα ασφάλειας μόνο είναι ζήτημα εσωτερικής αγοράς δεν μπορεί να έχεις μια ασφαλή εσωτερική αγορά αν δεν έχεις υψηλή ασφάλεια. ο πολίτης πρέπει να μπορεί να εμπιστεύεται ότι τα δεδομένα του δεν την χάνουν παράνομης εκμετάλλευσης ή εποπτείας. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Μπαίνω σε λεπτομέρειες και συγγνώμη γι' αυτό. Ένα άλλο σημείο. Είναι παράδοξο, όπως είπατε, κάποιες δομές δεν έχουν πρόσβαση σε 5G. Οι, οι, οι, διοκτικές αρχές, για παράδειγμα, μέχρι τώρα. η, η πρόσβαση δηλαδή σε 5G δεν μπορούσε να γίνει από τις, από τις ε, διοκτικές αρχές. Εμείς αυτό θα πρέπει να το υλοποιήσουμε τεχνικά, να μπορέσει δηλαδή να επιτρέψουμε στις διοκτικές αρχές να δουλέψουν αποτελεσματικά μέσα σε ένα περιβάλλον 5G. Σε συνεργασία και με τη Γενική Διεύθυνση Home και με τη Europol. Χρηματοδότηση. Μπορώ να σας δώσω κάποια πληροφορίες για τη χρηματοδότηση μέσω της γραμματείας. Το πρόγραμμα δράσης θέλει να έχει φιλοδοξία να υλοποιηθεί το δίκτυο 5G σε όλα τα κράτη-μέλη πριν το 2025. Προφανώς λόγω της γεωγραφικής διαφόρας, των γεωγραφικών διαιρέσεων, σε κάποιες χώρες θα είναι ταχύτερο από ό,τι σε άλλα. Εμείς προτείνουμε μια σειρά δράσεων για το ΣΕΦ2 με 3 δις για τη σύνδεση μεγάλο κομμάτι του οποίου θα πάει στην συνδεσιμότητα εκείνων των περιοχών της Ένωσης που χρειάζονται βοήθεια, είναι πίσω. Εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης, για παράδειγμα. Επίσης, πήγα πρόσφατα σε κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και της Βαλτικής. Ε, κάποια από τα πιο ασφαλή πλαίσια ασφάλειας που έχω δει είναι εκεί δεν πρέπει να ντρέπονται. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. Να πω και κάτι άλλο που άκουσα από κάποιους βουλευτές. Η Ευρώπη δεν ιστερεί στο 5G. Αν πιστέψετε την προπαγάνδα αυτή, θα πιστέψετε και άλλες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι σημαντικό. Τι θέλω να πω. Όπως σας είπα, δύο μεγάλοι προμηθευτές από τους τρεις είναι Ευρωπαίοι. Έχουν περίπου 35% όλων των ευρεσιτεχνιών στα 5G. Είναι σχεδόν στο 50% των βασικών διπλωμάτων. Δηλαδή αυτών που είναι οι δηλωθήσεις τεχνολογίες. Επιπλέον, αν δείτε τους τέσσερις κύριους φορείς και όχι τις μικρές, ε, τις μικρές επιχειρήσεις, έχουν 56% των ευρεσιτεχνιών ως προς την τεχνολογία. Είμαστε εκεί λόγω των προσπαθειών που κάνουν οι ερευνητικέ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και της βοήθειες στην έρευνα που δίνει η ΕΕ. Επίσης, δεν υπάρχει 5G. Κάποιες ανακοινώσεις προώθησης στην αγορά έχουν γίνει, αλλά δεν έχουμε πραγματικό 5G. Υπάρχουν, ας πούμε, γρήγορα, γρήγορες συνδέσεις στα σπίτια, στην, ε, στις ΗΠΑ που το λένε 5G, αλλά δεν είναι 5G. Του χρόνου θα ξεκινήσουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα πλήρες δίκτυο πέμπτης γενεάς που θα ολοκληρωθεί το 25. Μην αφήνετε να πείθεστε ότι το 5G έχει αρχίσει να ξεκινά. Αυτό που είπε ο κύριος Μπερτών είναι ότι στην θέση αυτή τεχνολογικής ηγεσία που έχουμε θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουμε ισχυρότεροι στην ανάπτυξη του, της έκτης γενεάς. Σας πήρα πολύ χρόνο. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλιώς να δώσω λεπτομέρειες στη γραμματεία για το τι θέλουμε να κάνουμε και στο πλαίσιο του νέου ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαβίνσκι. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ε, είπαν οι συνάδελφοι, ο συνάδελφος. Γιατί συνεργαζόμαστε πολύ και αυτό που είπα και στην ομιλία μου είναι τι κάνουμε για τις ε, στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις της ΚΕΠΑ σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις των κρατών μελών για τη χρήση της τεχνολογίας 5G και το ποιε είναι οι συνέπειε αυτών. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προετοιμάσει πολλά έγγραφα και έχουμε προετοιμαστεί ιδιαίτερω για την ασφάλεια για μας. Το 5G δίνει συνδεσιμότητα μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και πολλές λύσεις τελικά θα χορηγηθούν στους θα προσφερθούν στους καταναλωτές. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα του 5G και θα δοθεί δυνατότητα για τεχνητή νοημοσύνη και το δίκτυο λοιπόν αυτό ενέχει πολλούς, πιο πολύ, πολύ πιο πολλούς κινδύνους και πολλές πιο πολλές δυνατότητες ε, για κακόβουλους παράγοντες ε, εις βάρος των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερω εδώ και να τονίσω και την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ Έχουμε μια κινητική κήρυξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ και εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε τακτικέ συναντήσεις με τους ομολόγου μας στο ΝΑΤΟ αναφορικά με τα έγγραφα αυτά για την κυβερνοασφάλεια για να υπάρχει ένας ευρύτερο συντονισμό των δράσεων προκειμένου τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα κατά τον ίδιο τρόπο έναντι των κυβερνοεπιθέσεων και κυβερνοαπειλών. Έχουμε συναντήσεις σε επίπεδο αξιωματούχων, σε χαμηλό επίπεδο, για να καταρτήσουμε ε, πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, διάφορες ασκήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό. Το θέμα της κατάρτισης, λοιπόν, κρίσιμη σημασία, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να αντιλαμβάνεται πώς να απαντά σε τέτοιου είδους ε, απειλές. Κάποιοι δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι υπάρχει και κίνδυνος ε, στο σπίτι του το ίδιο. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική σκούπα έχει μικρόφωνο, έχει κάμερα και αυτό μπορεί να το επουλευλευτούν για συλλογή πληροφοριών, οποιοδήποτε κακόβουλος. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση των πολιτών, γιατί όλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς ε, αρνητικούς σκοπούς. Η συνεργασία λοιπόν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ είναι σημαντικό σκέλο και εδώ δραστηριοποιούμαστε έντονα. Και στην παρούσα φάση συναντηθήκαμε με τον Γενικό Επικεφαλή του ACA της Υπηρεσίας Επικοινωνίας του ΝΑΤΟ και μιλήσαμε για την πρωτοβουλία για 10.000 στρατιώτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα και προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο άλλο από το στρατιωτικό σκέλος να σας αναφέρω. Να επισημάνομαι ότι δεν μιλάμε μόνο για τον εξοπλισμό δικτύου. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με το διαδίκτυο των πραγμάτων για οτιδήποτε συνδέεται στο δίκτυο και οτιδήποτε θα μπορούσε εν δυνάμει να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τεθεί ένα σωστό πλαίσιο προκειμένου να αποφύγουμε την χρήση του εξοπλισμού αυτού. Ευχαριστώ, λέει ο Να ευχαριστήσουμε και τους δύο ομιλητέ μας που διευκρίνησαν τα πράγματα. Σα ευχαριστώ κύριε Ντόναχιου Ίσως είναι λίγο ασυνήθιστο το γεγονός ότι ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνατε. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Σαμπίνσκι. chers collègues, je vous propose... Προτείνω αγαπητοί συνάδελφοι να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, το σημείο που θα εξετάσουμε τη ημερήσιας διάταξης είναι αντιαλλαγή απόψεων για την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ. Συγγνώμη, είναι δύσκολο να με ακούτε και να σας ακούω γιατί υπάρχει θόρυβος. Παρακαλώ ησυχία. Έχουμε λοιπόν ε, τον κύριο Στέφανο ε, Τωμά, Διευθυντή για την ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΕΑΕ και τον κύριο Κόπολα, επικεφαλής των ε, επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακολουθήσαμε όλοι στενά τις πρόσφατες εξελίξεις, τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράκ, επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων, συγκεντρώσεις ε, διαμαρτυρίες εχθρικές έξω από την Αμερικανική πρισβεία, δολοφονία του στρατηγού Χαμενεή και απάντηση των Ιρανικών αρχών με ε, ε, την επίθεση εναντίον Αμερικανικών στόχων στο Ερμπίλ. Ε, το Ιράκ γίνεται, φαίνεται να γίνεται το νέο πεδίο μάχης, για αυτό το νέο επεισόδιο συγκρούσεων που διαφαίνονται στον ορίζοντα στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συγκρούσεις είναι σε σημείο αποφασιστικό, σε σημείο καμπής. Έχουμε αντιπαράθεση μεγάλη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωση σημαντικής, ε, ε, σημαντική κλιμάκωση και το Ιράκ είναι το βασικό ε, πεδίο όπου θα διαμηθούν όλα αυτά. Αυτά λοιπόν έχουν σχέση με την ικανότητα ανταπόκριση και δράση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και επιτόπου, αλλά και εντός των διαφόρων συμμαχιών και των εντός ΝΑΤΟ και εντός της συμμαχίας ενάντια του Νταές και ε, εντός του Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Ένωσης Ιράκ έχουμε ε, παρουσία ξένων στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράκ ε, και γενικά όλα αυτά τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Η υφιστάμενη κρίση Υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμώσει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και στο Ιράκ και στη Συρία ε, όλα αυτά ε, ήδη έχουν έρθει σε χειρότερη θέση λόγω των τουρκικών επιθέσεων στους Κούρδους στα βορειοναταλικά της Συρίας. Από εκεί και πέρα έχουμε ε, διαδηλώσεις στο Ιράκ και βίαιη καταστολή αυτών από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ και όλα αυτά δημιουργούν, μας εγείρουν διάφορα ερωτήματα. Σε ποιες συνθήκες λαμβάνει η χώρα η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Πριν δώσω το λόγο στου ειδικού τους, οι και να τους ευχαριστήσω βέβαια για άλλη μια φορά, θέλω να εκφράσω ε, μια, κάτι που με θλίβει και μια επιθυμία μου. Λυπούμε διότι ούτε ο προηγούμενος, ούτε ο τωρινός επικεφαλής ε, του UM Iraq δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα και επιθυμώ, εκφράζω την επιθυμία επικεφαλής των επιχειρήσεων της PSDC της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να έρχεται τακτικά, να μας κάνει έναν απολογισμό, να μας υποβάλει αναφορές στη δική μας υποεπιτροπή γιατί εμείς ασκούμε, ε, διαδραματίζουμε αυτό το ρόλο της άσκησης δημοκρατικού ελέγχου διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δημοκρατικά εκλεγέν και ασκεί αυτό το ρόλο του ελέγχου. Θα ήθελα λοιπόν να περάσετε αυτό το μήνυμα ότι είναι, προς το, ότι είναι συλλογικό το ενδιαφέρον των μελών της Επιτροπής μας να συναντηθούν με τους επικεφαλείς των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις να δώσω το λόγο στον κύριο Στέφανο Τομά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για την ευκαιρία που μου δίνετε στην παρουσίασή μου. Θα ήθελα να επικεντρωθώ, να εστιάσω το ενδιαφέρον μου στα βασικά στοιχεία ε, που αποτελούν τη στρατηγική αναθεώρηση και επισκόπηση της αποστολής μας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο μέλλον, αλλά και βασικά στοιχεία για τις ε, μελλοντικές προοπτικές μας. Και ε, θα παρουσιάσω λεπτομερώς την αποστολή και την διοίκηση που ασκούμε εκεί. Λοιπόν, η κατάσταση στο Ιράκ, η τωρινή, αυτή που βλέπουμε τώρα, δεν ήταν κάτι το απρόβλεπτο, δεν ήταν κάτι που δεν είχε κανείς προβλέψει. Ακόμα ε, και πριν υπάρξουν οι δυσκολίες για τις οποίες μιλήσατε κυρία Πρόεδρε και οι οποίες όντως τώρα υπάρχουν, είχαμε διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας, διαδηλώσει που απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα ενάντια στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Θα θυμάστε την παρέτηση του Πρωθυπουργού του Ιράκ τον Νοέμβριο του 2019. Άρα η κατάσταση είναι συγκεχημένη, είναι χαόδης, είναι περίπλοκη, είναι, όχι χαόδης, είναι φλού, συγκεχημένη και ε, περίπλοκη και αυτό έχει αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Αποστολή, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 κατόπιν αιτήματος των Ιρακινών αρχών και υπήρξε ενδιαφέρον να ε, προοδεύσουν στις μεταρρυθμίσεις του τομέα τους για την ασφάλεια και γι' αυτό ζήτησαν στρατηγική συμβουλευτική. Τα κράτη-μέλη θεώρησαν και αξιολόγησαν ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια τέτοια παρουσία. Η κατάσταση έχει αλλάξει βεβαίως με την πάροδο του χρόνου. Τώρα, διάφορα στοιχεία επηρεάζουν την προσπάθεια που καταβάλουμε εμείς οι Ευρωπαίοι εκεί. Χρειάστηκε πολύ μεγάλος χρόνος, πάρα πολύ χρόνος να διαμορφωθεί και να συγκροτηθεί η προηγούμενη Ιρακινή κυβέρνηση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, άλλοι παράγοντες, Popular Mobilization Forces. Είναι ένα περίπλοκο στοιχείο αυτό καθεαυτό. Τώρα, η αποστολή. Απαντά, αντιμετωπίζει αυτή την περιπλοκή κατάσταση στο Ιράκ με διάφορους τρόπους. Έχει να κάνει και με τις Ιρακινές αρχές, η δική μας αποστολή σε επίπεδο ΕΕ και προσπαθεί να προσαρμόζεται ε, στην τρέχουσα κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται. Άλλες πτυχές της αποστολής πρέπει να, πρέπει να τονιστούν. Ας πούμε, η αποστολή μας συντονίζει και κάνει το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων διεθνών παραγόντων και παικτών. Και αυτό είναι κάτι που κάνουμε και πρέπει να το τονίσουμε. Τώρα, τι μελιγενέστε και τι γίνεται. Είναι ακριβώς η στιγμή, θεωρούμε, κατά την οποία η παρουσία της Ευρωπαϊκή είναι, χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια η αποστολή μας, η Ευρωπαϊκή, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχέσεων, να καλλιεργήσει ένα δίκτυο σχέσεων και άρα θεωρείται και γίνεται αντιληπτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αξιόπιστος εταίρος. Εμάς μας βλέπουν διαφορετικά οι Ιρακινοί ομόλογοι μας σε σχέση με τις μη ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε ο ουδέτερος συνομιλητής σε σχέση με τους άλλους παίκτες και αυτό το στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι μας αντιλαμβάνονται. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που διαμορφώνουν ε, τη θέση μας. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, η παρουσία της UAM είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα της χώρας αυτής καθεαυτής. Μόνο με την παρουσία μιας ορατής δύναμης ασφαλείας, αποστολής ασφαλείας στην περιοχή και με την απλή παρουσία το ότι είναι αυτή ορατή, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ε, στους ομολόγους μας, ότι έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη και τη δέσμευση για την διατήρηση της σταθερότητας. Άρα, με τα κρατημέλη έχουμε καταλήξει το εξή συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή είναι απαραίτητη, είναι σημαντική, πρέπει να παραμείνει και οι αλλαγέ που σημειώνονται στο Ιράκ οι οποίες ε, δεν είναι, δεν είναι ενδογενείς, οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες κατά κύριο λόγο, διότι το Ιράκ είναι η χώρα και η επικράτεια όπου ε, συγκρούονται οι περιφερειακές δυναμικές και βρίσκουν ε, το ξέσπασμα σε αυτή τη συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια. Επομένως πρέπει να είμαστε παρόντες για να εγγυηθούμε την μελλοντική σταθερότητα στη χώρα. Και με αυτά να δώσω το λόγο στον στρατηγό Κόπολα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής και τους βουλευτές. Να ξεκινήσω. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη αναφέρθηκαν για την κατάσταση στη ασφαλεία στο Ιράκ μετά τον, τη δολοφονία του κυρίου Σουλεϊμανή. Να πω απλώς ότι η αποστολή μας στο Ιράκ συνεχίζει να λειτουργεί παρότι το περιβάλλον ασφάλειας και το πολιτικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολα. Οι ενδογενείς αδυναμίες του Ιράκ και η ανάγκη παγίωσης ε, των θεσμών ε, για να παράσχουν ασφάλεια στους πολίτες είναι μια προσπάθεια μακράς πνοής για την Ένωση και για την συμβουλευτική αποστολή μας. Να κάνω μια παρατήρηση τώρα. Σε μια συνάντηση που είχε ο οριστής ε, επικεφαλής αποστολής ε, στο Ιράκ με τον πρέσβη του Ιράκ εδώ την περασμένη εβδομάδα έγινε σαφής διάκριση μεταξύ των ξένων δυνάμεων που σύμφωνα με το ψήφισμα του Ιρακινού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα και της αποστολής της ε, Ένωσης. Η αποστολή μας αναγνωρίζεται ως κάτι διαφορετικό, αυτό το λέω εξ αρχής. Η EUAM είναι μια μη εκτελεστική αποστολή ε, διαχείρισης κρίσεων με πολίτες στα πλαίσια της ε, ΚΕΠΑ. Παρέχει στρατηγική συμβουλευτική στην κυβέρνηση στη Βαγδάτη για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης ε, των τόσο αστικών, τόσο πολιτικών και όσο και στρατιωτικών δομών. Δεν παρέχουμε εξοπλισμό, δεν παρέχουμε κατάρτιση όπως κάνουμε αλλού παρότι συντονίζει στενά τις προσπάθειες με τους εταίρους που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Η αποστολή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017. Είναι η νεότερη δηλαδή αποστολή, περιμένοντας την πλήρη ανάπτυξη της αποστολής μας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. ενισχύσαμε την παρουσία μας στη χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα, αναπτυσσόμαστε, έχουμε αλλάξει σημαντικά ήδη, 60 άτομα είναι πλέον, διπλασιάστηκε δηλαδή ο αριθμός των, ε, των, των μελών της αποστολής. Μέχρι τώρα η αποστολή έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία της ως βασικό εταίρο της ε, ρακινή πλευράς, παρέχει συμβουλευτική σε πολλά επίπεδα, διοικητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα ζητήματα ασφάλειας, για την εφαρμογή με κανονικό τρόπο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πέραν της Εθνικής Στρατηγικής για την Ασφάλεια και της Στρατηγικής κατά τη, του φονταμεταλισμού, του εξτρεμισμού και, τη, το, της τρομοκρατίας. Ε, παρέχει συμβουλευτική για εξυπνότερη αστυνόμευση και κατάφερε να οργανώσει και να θεσπίσει την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δομών ενοποιημένης ε, διαχείρισης των συνόρων της χώρας και της Frontex στη Βαρσοβία. έχουμε πολλούς τομείς που προχωράνε. Στην αποστολή συνεργαζόμαστε στενά με την αντιπροσωπεία της Ένωσης για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλει εκεί η Ένωση και με τα κράτη-μέλη βέβαια. Θέλουμε να ενισχύσουμε την συνοχή της δράσης της Ένωσης ε, στο πλαίσιο αυτό. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Υποστηρίζουμε, όπως είπα, μακροχρόνιες διαδρασίες Αλλά θέλω να λύσω και κάποιες πρόσφατες, ε, κάποια πρόσφατα επιτεύγματα. Όταν οι δυνάμεις της χώρας έδειξαν αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις ε, πρόσφατες ε, διαδηλώσεις, προσπαθήσαμε να τους παράσχουμε πληροφορίες για το πώς γινόταν αυτό σε άλλες χώρες, παρέχοντας αναλογική μορφή λειτουργίας. Ταυτόχρονα ετοιμάσα μια σειρά συνεδριάσεων ε, σε πλατφόρμας και στη Βαγδάτη και στο Έρμπιλ για να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων μειονοτήτων της χώρας, του Υπουργείου και των δικαστικών. Η υποστολή υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ιράκ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέρος της συνεργασίας της με τον ΟΗΕ και την Europol. Κάτι κρίσιμο για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως είπα νωρίτερα. Διευκόλυνε την ε, συνεργασία μεταξύ της Frontex και των συνοριοφυλάκων της χώρας. Τώρα, η μεταρρύθμιση του κλάδου για να σέβεται περισσότερο το κράτος δικαίου. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, μια μεγάλη πρόκληση που επιδεινώνεται από την επιδείνωση της ασφάλειας. Η αποστολή θέλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, θα πω σε λίγο κάτι γι' αυτό, και την αύξηση της έντασης επιτόπου. Πολιτικά, η παρέτηση του Πρωθυπουργού του Ιράκ το Νοέμβριο υποχρέωσε την αποστολή να δημιουργήσει νέες σχέσεις με βάση την εμπιστοσύνη και την αμοιβή εμπιστοσύνη μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι εταίροι μας, ε, οι αντισυμβαλόμενοι στο Ιράκ, ε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν έδειξαν πάντα ενδιαφέρον ε, συνεργασίας μαζί μας και χρειάστηκε να δουλέψουμε στενά για να τους πείσουμε για την χρησιμότητα της παρέμβασής μας. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συμβουλευτική για ζητήματα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, προώθηση καλύτερης λογοδοσίας, ε, ε, μηχανισμούς ε, παρακολούθησης από τους πολίτες. Η εμπλοκή της Ένωσης με την κοινωνία των πολιτών ενισχύεται. Βρίσκουμε τρόπους για την υποστήριξη της ασφάλειας σε πιο, αποτελεσμα, με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Βεβαίως, οι προκλήσεις παραμένουν πολλές, έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που πήραν μπρος με τον αγώνα κατά του Ντάες. Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά τον Ιανουάριο. Με... Εμείς έχουμε ένα προσωπικό 60 τόνων, 20 είναι, ε, ήταν εκεί την περίοδο εκείνη. Δεν γύρισαν οι περισσότεροι στο Ιράκ μετά τον Ιανουάριο με δική μου εισήγηση. Θα επιστρέψουν μετά την δική μου επίσκεψη στο Ιράκ, πάω εκεί την Δευτέρα και τότε θα αποφασίσω αν θα επιστρέψει περισσότερο προσωπικό στη χώρα για να ξεκινήσουν ε, την συνεργασία εκ νέου με τις τοπικές αρχές και θα δω και τον Υπουργό Εσωτερικών παρεμπιπτόντως. Για ένα διάστημα η, η αποστολή δεν μπορούσε να ταξιδέψει έξω από τη Βαγδάτη. Έχουμε δύο σημεία μέσα στο... δύο, δύο ε, στην, πράσινη, στην παλιά πράσινη ζώνη και στην παλιά κόκκινη ζώνη που είναι πιο κοντά στην, ε, στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα μπορούμε να ταξιδέψουν, να ταξιδέψουν εκτός της, ε, του χώρου τους για επιχειρησιακούς λόγους για να μπορέσει να πάει και στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου υπάρχει κοινό επιχειρησιακό κέντρο και αποτελεί τη βάση μας στο Υπουργείο Εσωτερικών που χρησιμοποιούμε για συναντήσεις, κατάρτιση, όχι κατάρτιση, συμβουλή δηλαδή, υπαρχή συμβουλευτικής. ή για να κάνουμε συντονισμό με άλλες αρχές, εθνικές ή διεθνείς. Η κατάσταση συνολικά είναι σταθερή. Δεν υπήρξε επίθεση εναντίον μας. Καμία επίθεση δεν έγινε δίπλα στις ε, ε, εγκαταστάσεις μας. Δεν επηρέασαν ε, τις ε, δραστηριότητές μας. Μετά την επισκεψή μου την Δευτέρα είμαι βέβαιος ότι θα επανεξετάσουμε κάποια από τα μέτρα που έχουμε λάβει για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Δεν περιμένω να γυρίσει όλη η αποστολή επιτόπου, αλλά σίγουρα μπορούμε να αυξήσουμε την παρουσία μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας και την υποστήριξη προς τις τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στον γύρο των ερωτήσεων και να ξεκινήσουμε από πλευρά των Πρασίνων με την κυρία Νόημαν. Ευχαριστώ. Κύριε Τον Κυρικόπολα, έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Είπατε ότι η αποστολή αυξήθηκε με προσωπικό 60 ατόμων επιτόπου από την αναθεώρηση της προηγούμενης εντολής πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε νομίζω ότι έχουμε βρει τρεις τάσεις, ε, διαπιστώσει τρεις στάσεις στο Ιράκ, ανησυχητικές. Καταρχάς η αποστολή αυτή, όπως είπατε, είναι για μια μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας του Υπουργείου Ιστορικών. Εκ παραλίλου, βλέπουμε ε, ε, φορεί τη κυβέρνηση στο Ιράκ να πυροβολούν διαδηλωτέ στου δρόμου χωρί καμία αμερόληπτη έρευνα. Και πρέπει να σα πω ότι ήταν πολύ έντονη η διατύπωση των ε, γεγονότων. Τι τάσει λοιπόν είναι αυτέ Αν ε, εκπαιδεύουμε την αστυνομία και εκ παραλίλου έχουμε ε, την αστυνοφνουρά πολιτοφυλακή η οποία βγαίνει στους δρόμους και κάνει το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι κάνει. Ύστερα, να δούμε ε, Πώ γίνονται αντιληπτοί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρούνται ε, αμερόληπτοι οι φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την διευκόλυνση τη συζήτηση μεταξύ τη κυβέρνηση και των διατελετών. Δεν έχω δει όμως μεγάλη δράση προ την κατεύθυνση αυτή και ύστερα η δολοφονία του Σουλεμανή στο Ιράκ το οποίο ε, φέρνει όλου του ανθρώπου αυτού, το προσωπικό αυτό, σε πολύ ευάλωτη θέση. Αναρωτιόμαστε κατά πόσον είναι επιθυμητή η παρουσία του εκεί. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ε, ενισχυθεί η παρουσία μας στο Ιράκ. Είναι πολύ βασικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνει τις προσπάθειές της και σε μη στρατιωτικό επίπεδο. Δεδομένου λοιπόν όλων αυτών των εξελίξεων των τελευταίων μηνών και δεδομένου του ότι η εντολή είναι υπό αναθεώρηση, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η εντολή για να εσημειθούν σημαντικές αλλαγές επί τόπου και αν δεν μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αλλάξουν την εντολή αυτή, έχει κανένα νόημα να συνεχίσουμε με 60 άτομα δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση επίσης, δεδομένου του διχασμού της ε, ε, κοινωνίας των ε, Ιρακινών, της κοινότητας και Σουνιτών και δεδομένου ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας θα πρέπει να αποτυπώνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται λεπτές από όλο τον κόσμο ως έχουν Δεν ξέρω τι ποσοστό ε, εκπροσώπησης υπάρχει συνειδητών και Σεϊτών στις δυνάμεις αυτές, 60-40% αλλά τμήμα της προσπάθειας μεταρρύθμισης είναι να τους πείσουμε ότι προκειμένου να οικοδομηθεί ένα κράτος από κοινού θα πρέπει και στους ευαίσθητους, ευάλωτους τομείς όπως στις δυνάμεις ασφαλείας, στην αστυνομία να υπάρχει η σύνθεση αυτή που θα αποτυπώνει και τη σύνθεση του πληθυσμού. Ο πρέσβης μας δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται η μη στρατιωτικές μα δυνάμει, Αυτό είναι καλό. Διευκρινίστε όμως, παρακαλώ. Είναι σαφέ κατά πόσον η κυβέρνηση θα ακολουθήσει επιτέλου τις συστάσεις του Κοινοβουλίου ή όχι. Και αυτή η έκκληση για τι αμερικανικέ δυνάμει να καταρτήσουν ένα σχέδιο αποχώρηση έχει αποσταλεί και στις δικές μας δυνάμει. Πώς έχουν τα πράγματα Ποιε είναι οι πιο πρόσφατες εξελίξει στο κουρδικό τμήμα. Είπατε ότι υπάρχουν και άτομα στο Ερμπίλ. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο εύκολα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τι αρχές. Καταρχάς γιατί είναι ειρηνική ως επιτοπλίστων η κατάσταση και επειδή δεν υπάρχει το πρόβλημα των δύο κοινοτήτων το οποίο εντείνει α, τα προβλήματα και τι τριβέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κίτσος. Thank you. Ευχαριστώ. Κάποιε ερωτήσει έχω να θέσω γιατί προσπαθώ να κατανοήσω τι ακριβώ συμβαίνει στο Ιράκ. Όσο υπονομεύεται η κατάσταση στο Ιράκ, το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία, τόσο πιο έντονο γίνεται το πρόβλημα το μεταναστευτικό στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, εξ όσων γνωρίζω, το Ιράκ είναι η μεγαλύτερη, δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγέα ε, πετρελαίου ανάμεσα στα κράτη ΟΠΕΚ. Και από ό,τι βλέπω έχουμε 5 εκατομμύρια βαρέλια α, κάθε ημέρα. Τεράστιες ποσότητες. Και φυσικά τεράστιο ποσό χρημάτων. Πώς εξηγείται λοιπόν το γεγονός ε, ότι βρίσκονται σε τόσο δεινή οικονομική κατάσταση ο λαός του Ιράκ. Υπάρχουν λοιπόν τόσο πολλά χρήματα. Είναι θέμα διαφθοράς της κυβέρνησης, είναι θέμα των πολυεθνικών ομήλων και των συμφερόντων τους. Ποια είναι η άποψή σας. Δεύτερη ερώτηση. Τι πρόκειται να γίνει στο Ιράκ. Φυσικά και υπάρχουν εντάσει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων πολιτειών. Οι Σιήτες ε, είναι η πιο ισχυρή δύναμη και στην εθνοφρουρά και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά παράλληλα οι διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα τους προηγούμενους μήνες και από ό,τι διάβασα και σήμερα στους Financial Times ε, είναι όλο και πιο εκτενείς ε, προς την Πάσρα νομίζω πάνε έχουν να κάνουν κυρίως με ένα τμήμα της κοινωνίας στο Ιράκ που δεν θέλει να συνδεθεί με το πολιτικό σύστημα και με τον ανταγωνισμό μεταξύ Ισίτων και Σουνιτών. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της κοινωνίας, αυτοί οι διαδηλωτέ που καταπιέζονται από τις κυβερνητικές δυνάμεις και είναι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες στον αριθμό. Έχουν οποιαδήποτε ευκαιρία. Μιλάμε για πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και τέλος, τι γίνεται με την ε, στρατηγική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουν ε, ε, πάει στο Κουβέιτ για να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Ενημερώστε μας αν θέλετε. Δώστε μας πιο πολλά στοιχεία. Ευχαριστώ ο κύριος Κρίς Πέιταρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν χθες. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Μπέρικα ε, από το ΝΑΤΟ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακούσαμε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Τι θα γίνει με την ανακοίνωση του Πρόεδρου του, τον ΗΠΑ για τη μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είμαστε σε φάση έντονων συζητήσεων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το ΝΑΤΟ θα δραστηριοποιηθεί πιο έντονα σε σχέση με το παρελθόν, όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Ρωτώ λοιπόν, καταρχάς, έχετε λάβει και εσείς αυτή την πληροφορία. Κατά δεύτερον, αν ε, όντω έχετε λάβει τις πληροφορίες αυτές, ε, αν τις έχετε λάβει κρίμα, αν τις έχετε λάβει όμως τις πληροφορίες αυτές, για πείτε μας τι πιστεύετε γι' αυτό. Και τρίτον, ποια θα είναι η επίδραση σε αυτά που κάνετε εσείς, που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ όντω δραστηριοποιηθεί πιο έντονα εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρι. Η ερώτησή μου προς τον ε, στρατηγό τον κύριο Κόπουλα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σα. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Καταρχά, επιβεβαιώνεται ότι η αποστολή στην παρούσα φάση βρίσκεται σε stand-by. Κατά δεύτερον, τι μέτρα ασφάλεια, αν μπορείτε να τα συζητήσετε, έχετε για το προσωπικό που βρίσκεται στο Ιράκ. Τι αναγκαστήκατε να λάβετε ως μέτρα δηλαδή ασφάλειας και κατά τρίτον, αντιλαμβάνεστε διαφορές στις συνομιλίες σας με τους ε, Ιρακινούς ε, ομολόγους σε ό,τι αφορά μια διαφορετική αντίληψη πλέον μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνονται αντιληπτές αυτές οι δύο δυνάμεις. Ο κ. Thank you. I will... Ευχαριστώ και θα μιλήσω ελληνικά. Uh, νομίζουμε ότι πλέον τα παραδείγματα δεν είναι, δεν είναι μοναδικό το παράδειγμα του Ιράκ για να βγάλουμε συμπέρασμα. Είναι και η Συρία, είναι και η Λιβύη. Μιλάμε για πολύχρονες ε, για πολύχρονη εισβολή, κατοχή, βομβαρδισμοί, εμφύλιες διαμάχες και πρέπει να βγει συμπέρασμα από όλη αυτή την πρακτική που ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Και ο πυρήνας θεωρώ τον... Ε, εξελίξεων είναι ακριβώς το ζήτημα του τερματισμού της κατοχής. Αυτό είναι ο πυρήνα των εξελίξεων που οδηγούν αυτή τη στιγμή στο Ιράκ πρώτον και το δεύτερο στοιχείο είναι ποιος θα επωφεληθεί από τον όποιο τερματισμό ή όποια διαφορετική διαδικασία μετάβασης την επόμενη μέρα. Και επειδή σε αυτές τις εξελίξεις έχει κομβικό ρόλο ο έλεγχος του στρατού, θα θέλαμε τη γνώμη σας για το ποιος αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι, ποιος ελέγχει το στρατό σε σχέση και με την κατάσταση και που έχει διαμορφωθεί με την αντιπαράθεση με το Ιράν που στο επίκεντρό του έχει την σωμάτωση των λεγόμενων ε, ομάδων αυτών ε, λαϊκής κινητοποίησης που ε, έχουν ε, ρόλο στις, σε σχέση με το στρατιωτικό συσχετισμό στη χώρα. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστώ από την New Europe. Ο Σας ευχαριστώ. Και φαντάζομαι ότι μία από τις εξελίξεις ε, για το Ιράκ που επηρεάζουν εδώ και την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια είναι οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ISIS και τις άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό είναι προφανές και ατυχές ότι τα περιστατικά του φετινού έτους και η μάχη κατά της ε, ISIS στην ε, επικράτη του Ιράκ και προφανώς αυτό συνδέεται και με τα τεκτενόμενα στη Συρία. Όλα αυτά λοιπόν θα αποδυναμωθούν αυτές οι μάχες. Θα θέλαμε να ακούσουμε λοιπόν και από δική σας πλευράς πώς ε, αντιλαμβάνεστε τις ε, περαιτέρω τρομοκρατικές, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες στο Ιράκ, με την ευρωπαϊκή παρουσία, με παρουσία άλλων δυνάμεων. Τι ζημιά προκάλεσαν τα γεγονότα της αρχής του έτους και οι ενδεχόμενες συνέπειες στο άμεσο μέλλον αλλά και πιο μακροχρόνια από στρατηγικής άποψης. Ευχαριστώ. Η κυρία Σκίτεντόλα ήρθε η επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Ιράκ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία Σκίτενταλ. Ευχαριστώ πολύ και θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Καθυστέρησα. Ήμουν στην Επιτροπή Απασχόλησης, όπου έγινε παρουσίαση της ε, έκθεσής μου γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να είμαστε παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ. Πρόεδρε, χαίρομαι. Και είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Και για να περάσω στο μήνυμα που έχω να σας δώσω προς την Επιτροπή σας σήμερα. Είδαμε ότι το ψήφισμα του Ρακινού Κοινοβουλίου, το οποίο εκτίθηκε ε, ω επιτοπλίστων από αποσύτε βουλευτέ για την αποκάλυψη ξένων δυνάμεων μέσα στη χώρα, είναι κάτι πολύ αρνητικό σε εξέλιξη. Και αν όντω περάσει, προφανώ θα αποτρέψει ε, τους διεθνεί εταίρου ε, που πολεμούν το Ισλαμικό κράτος και υπονομεύει τη δυνατότητά τους να πετύχουν τους στόχους τους. Όπως τα γνωρίζετε, η Σουηδία είναι από τις χώρες εκείνες που έχει στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ και η στρατιωτική επιχείρηση περιλαμβάνει περίπου 70 στρατιωτικούς που ο σκοπό έχουν να εκπαιδεύουν και να συμβουλεύουν τις δυνάμεις του Ιράκ στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους. Δεν έχει τελειώσει αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος ακόμα και είμαστε 30 χιλιόμετρα ε, έξω από τη Βαγδάτη μια βάση η οποία έχει αποτελέσει ε, έχει δεχτεί επιθέσεις σε διάφορες ε, περιστάσεις μετά την τηλεφωνία του Σουλημανή. Και εδώ να υπογραμμίσω ότι η απόσυρση δυνάμεων από το Ιράκ αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο έλεγχο των Ιρανικών, της Ιρανικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες τριβές και αυτό θα οδηγήσει σε άνοδο πάλι των Ισλαμικών ε, δυνάμεων του Ισλαμικού κράτους και θα αποτελέσει μεγάλη απειλή για την ε, κυριαρχία του Ιράκ. Τα αποτελέσματα της ε, συμβουλευτικής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας του Ιράκ έχουν τεράστιες επιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει αρρωγή και υποστήριξη στις Ιρακινές δυνάμεις για τις ε, πρακτικές αυτές. Μόνο οι κρατικοί φορείς είναι σε θέση να επιβάλλουν τη σταθεροποίηση, να προχωρήσουν την εξέλιξη και να αποτρέψουν περαιτέρω σειράξεις. Μόνο έτσι λοιπόν η χώρα θα μπορέσει να κάνει την πλήρη μετάβαση σε μια ευρυθμή δημοκρατία. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ιράκ σε συνεργασία με τις ε, αρμόδιες επιτροπέ θα συνεχίσει προφανώ να παρακολουθεί στενά τι εξελίξει τη κατάσταση ασφαλεία στο Ιράκ και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συνεργασία με την Επιτροπή σα. Και καλώ του συναδέλφου σε μια συνάντηση η οποία θα λάβει χώρα 31 Ιανουαρίου με εκπροσώπους του Ιράν και της Αραβικής Χερσονήσου για να εξετάσουμε την κατάσταση στο Ιράκ και στην ε, Μέση Ανατολή εν γέννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και το λέω τώρα έχει ο κύριο Στομά και ο στρατηγό κ. Κοπολά. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα διάφορα ερωτήματα που μου θέσατε. Σίγουρα ορισμένα από τα ερωτήματα αναφέρονται σε θέματα που ξεπερνούν τις δικές μας αρμοδιότητες, όμως επιτρέψτε μου να σχολιάσω και να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια από αυτά. Πώς μας αντιλαμβάνεται το ευρύ κοινό, την UAM, τη στηρίζει, την ανέχεται, το ότι εμείς ανεχόμαστε, εν πάση περιπτώσει, την απάντηση των Ιρακινών αρχών στις διαμαρτυρίες. Κοιτάξτε, η αποστολή μας συμβουλεύει σε στρατηγικό επίπεδο. Στηρίζουμε την τήρηση το, και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά για να γίνουν αυτά σεβαστά πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα και στηρίζουμε τη δημιουργία αυτής της κουλτούρας στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλου του πλέγματος. Η παρουσία της αποστολής σε στρατηγικό επίπεδο εντός των δομών ασφαλείας στο Ιράκ είναι ένα στοιχείο το που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει, να μαθαίνουμε τι συμβαίνει. Και έμεσα είναι ένα στοιχείο ελέγχου και προειδοποίησης. Η παρουσία της αποστολής είναι ένας παράγοντας που κάνει την Ιρακινή απάντηση να είναι πιο προσεκτική ενδεχομένως. Και αυτό έχω να πω για αυτό το θέμα. Τώρα, είμαστε ικανοί να φέρουμε αποτελέσματα με βάση την εντολή μας, από τη στιγμή που η κατάσταση είναι συγκεχημένη και περίπλοκη. Κοιτάξτε, η στρατηγική αναθεώρηση που παρουσιάζουμε δίνει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Υπό ποια έννοια. Θέλουμε να ασχοληθούμε με θέματα τα οποία σε στρατηγικό επίπεδο επηρεάζουν την ικανότητα των δυνάμεων ασφαλείας να είναι αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιμείνουμε σε θέματα όπως η διαχείριση συνόρων, ε, θέματα αντιτρομοκρατίας, αντιτρομοκρατικής. Γίνεται συζήτηση για περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος των ανθρωπίνων πόρων και της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Με ποιο σκοπό θα πείτε. Είναι απαραίτητο αυτό, απαντώ. Για παράδειγμα στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Στον εντοπισμό του πού είναι οι δυνάμεις και ποιες είναι οι δυνάμεις κάθε φορά που υπάρχει κάποιο ε, σημείο τριβής. Ορισμένοι τώρα αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή τους το πρόβλημα της πρόσβασης. Ποιο αντίκτυπο τελικά έχουμε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον Ιρακινό λαό. Έχουμε περιορισμένη πρόσβαση, είναι η απάντηση. Το είπα και στην παρουσίασή μου. Ο συνάμα όμως αυτό μας επιτρέπει να εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε θέματα που μας απασχολούν περισσότερο στο μέλλον, που θα μας απασχολήσουν περισσότερο στο μέλλον. Για παράδειγμα, η αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού είναι ένα τομέα πάνω στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ε, με τους Ιρακινούς ομολόγους, κάτι το οποίο θα αποτελέσει, θα καταστεί ευεργετικό και για μας και για εκείνους. Μιλήσατε και για το Ερμπίλ. Το Ερμπίλ είναι μια άλλη πτυχή της ε, σκέψης μας αυτή τη στιγμή και πτώμαστε να ανοίξουμε εκεί γραφεία και άρα θα έχουμε μεγαλύτερο μοχλό, αν θέλετε, τοπικά, δυνατότερο και θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί και στη Βαγδάτη και να έχει επικοινωνία με τις Ιράκινες αρχές. Είναι μια ευκαιρία, το σκεφτόμαστε. Τώρα για το ΝΑΤΟ. Η αποστολή συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, γίνεται συντονισμός με τη σχετική νατοϊκή αποστολή στο Ιράκ και είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο γιατί η συνεργασία έχει να κάνει και με θέματα διαφάνειας, με θέματα φορητότητας, κινητικότητας, με θέματα φύλου, διάστασης των δύο φύλων. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις ικανότητες των Ιρακινών δυνάμεων, αλλά και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εμείς και βλέπουμε τα πράγματα. Δύο δευτερόλεπτα επιτρέψτε μου να σταθώ στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το ε, ανέφερε και ο κύριος Κόπολα. Ξέρω ότι φαίνεται ίσονος σημασία ή άσχετο με βάση την επίγουσα κατάσταση, αλλά για μας είναι σημαντικό πρώτη αποστολή που περιλαμβάνει ε, ε, ε, ρητή αναφορά στο θέμα στην περιγραφή της εντολής της. Άλλωστε, η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών ομάδων παγκοσμίω. Και επίσης, κάτι το ενδιαφέρον είναι το εξή. Η Ιρακινή είναι διαιρεμένη σε πολλά επίπεδα, π.χ. σε θρησκευτικό επίπεδο. Όλοι όμως θεωρούν αυτούς απογόνους του αρχαίου πολιτισμού των Βαβυλωνίων και των Ασσύριων και ούτω καθεξής. Άρα η πολιτιστική κληρονομιά τι είναι να τους ενώνει και να μειώνει ε, τις διαιρέσεις και τους διχασμούς και τις διχόνοιες. Είναι ιδιαίτερο αυτό το ζήτημα και μπορεί να μας βοηθήσει για να καλλιεργήσουμε σχέσεις και δεσμούς μεταξύ ε, των διαφόρων κοινοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο Στρατηγός Κόπελα παρακαλώ. Ευχαριστώ Στέφανο. Συμφωνώ απολύτως. Ε, με τον Στέφανο, διαφυσβήτητα, συμφωνούμε 100%. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ περισσότερο στα ερωτήματα που μου απευθύνατε προσωπικά στην αρχή. Ε, μπορεί να τα καταφέρει μια αποστολή των 60. 30 είμαστε στην αρχή. Να, να τροποποιήσει δραματικά το τομέα της ασφάλειας στο Ιράκ. Η απάντηση είναι όχι, όχι σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Αλλά είμαστε εκεί. Είμαστε παρόντες, στέλνουμε τα μηνύματά μας, συνεχώς δεν σταματούμε να κυνηγάμε την ανώτατη Ιρακινή διοίκηση και να την πλημμυρίσουμε με τα μηνύματά μας για να τις περάσουμε τα σωστά μηνύματα όπως θα θεωρούμε εμείς. Έχουμε εντολή και η εντολή είναι να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικό επίπεδο σε μια χώρα κατά την οποία οι αστυνομικέ δυνάμει υποτίθεται είναι 600.000 άνθρωποι, αλλά αν ρωτήσει του επικεφαλεί του ποιοι είναι αυτοί και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουν. Δεν έχουν ικανότητα ελέγχου και διαχείριση των αστυνομικών του αρχών και του πληθυσμού τους, ε, του αστυνομικού. Ε, οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν ένα περίπλοκο σύστημα βάσης δεδομένων για, για, τη διαχείριση των ανθρωπίνων στο πόρων. Μπορεί να το πληρώσουν, αλλά προς το παρόν οι Ιρακινοί δεν θα είναι σε θέση να το χειριστούν αυτό το σύστημα ε, με τη βάση δεδομένων, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Και προσπαθούμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι διμερές το project αυτό, και απαντώ και στο ερώτημα για τη συνεργασία που έχουμε με τους Αμερικανούς, να ένα παράδειγμα, δηλαδή τις τεχνικές ικανότητες των Αμερικανών προσπαθούμε να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες της αστυνομία για να μπορούν να ελέγχουν το προσωπικό τους, να ξέρουν που βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε συντονισμό και με τον ΝΑΤΟ και με τη Συμμαχία και με Κάθε φορά που είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί συντονιστικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι συντονίζονται μαζί μας, αλλά αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Τώρα, αν θα κάνουμε τη διαφορά αύριο, όχι, όχι, δεν θα υπάρξει διαφορά αύριο, σα το λέω, αλλά πρέπει να επιμείνουμε, να παραμείνουμε εκεί παρόντες. Ήμασταν 30, καταφέραμε να γίνουμε 60, θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερη και ισχυρότερη εντολή, όσο περισσότερο καταλαβαίνουν τα κράτη-μέλη τι θέλουν από το Ιράκ και τι θέλουν να κάνουν με το Ιράκ. Εμείς είμαστε εκεί και προσαρμοζόμαστε στην κατάσταση. Ήμασταν Είχαμε εμπλακεί πολύ στο θέμα της αστυνόμευσης των διαδηλώσεων και των πόριών. Μετά είχαμε τα προβλήματα του Ιανουαρίου και χρειάστηκε να σταματήσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία μαζί τους και να τους μιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Έχουμε μειωμένη παρουσία επιτόπου και αυτό είναι προσωπική μου ευθύνη, αν θέλετε, αρμοδιότητα. Να καλέσω και τους 60 και να τους πω επιστρέψτε στο Ιράκ μπορώ να το κάνω, αλλά πριν το κάνω θέλω να πάω και να δω τι γίνεται και να δουλέψω με τους ανθρώπους επί τόπου για να καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει διέξοδος, δεν μπορούμε να φύγουμε από εκεί ξεκινήσαμε πριν από δύο ε, χρόνια με μια εντολή όχι τόσο φιλόδοξη, πράγματι. Την αναθεωρήσαμε την εντολή, αυξήσαμε την ευρωπαϊκή παρουσία και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσουμε με αυτό το σκεπτικό σε βάθος χρόνου και ενδεχομένως σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να έχουμε περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη και πιο ευρεία εντολή. Είναι όμως πράγματα που θα εξεταστούν σε βάθος χρόνου, με την πάροδο του χρόνου, σε εύθετο χρόνο μάλλον. Το γεγονός ότι Ήδη έχουμε κάνει το γύρο της χώρας και έχουμε επισκεφθεί και άλλες περιοχές και περιφέρειες, όχι μόνο στο Ερμπίλ. Έχουμε συνομιλήσει με τοπικούς επικεφαλείς των αστυνομικών αρχών και όλοι μας λένε στηρίξτε μας. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε το οποίο ήταν ε, ε, ευνοϊκό και μας είπε επεκταθείτε στο Ερμπίλ. Να δούμε αν, και πότε θα το καταφέρουμε. Και το ίδιο θα κάνουμε όπως και στην αποστολή με την Ουκρανία ή αλλού. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, η αποστολή μα είναι παρούσα σε τέσσερα διαφορετικά σημεία γεωγραφικά πέραν του Κιέβου και εκτός από το Κίεβο. Δηλαδή είναι μια εξελεκτική διαδικασία η οποία αλλάζει. εκτος απο το κιβο δηλαδη ειναι μια προσέγγιση ενεργητική ε, για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ε, πάντοτε μπορούμε να προσαρμοζόμαστε με την κατάσταση και αυτούς τους λίγους πόρους που έχουμε να τους εφηρώνουμε στους τομείς και στους κλάδους όπου θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Αν πιστεύουμε ότι σε ένα τομέα δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα ιδιαίτερο, π.χ. στην αντιτρομοκρατική δράση, τότε το αφήνουμε αυτό κατά μέρο και επικεντρωνόμαστε σε άλλους τομείς όπου μπορούμε κάποια πράγματα να πετύχουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ας είμαστε ειλικρινείς. 60 ανθρώπους έχουμε μόνο επί τόπου και 60 δεν είναι η σύμβουλη, είναι η αποστολή με, το, με τον επικεφαλής για την ασφάλεια, τον αρμόδιο για τις επικοινωνίες, τον αρμόδιο για τον εφοδιασμό, την ε, επιμελητία και ούτω καθεξής. 60, 60 είναι το συνολικό νούμερο. Δηλαδή και το διοικητικό προσωπικό υποστήριξης πέραν των συμβούλων. Δεν υπάρχει τρόπος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Ή μάλλον ναι, υπάρχει. Τι θέλουμε να πετύχουμε. Ποια είναι η εντολή. Ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράκ. Ανάλογα με την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, μπορώ να σας πω ότι χρειαζόμαστε 60 ή 600 ή 6.000 ή 60.000. Δεν είναι μικρή χώρα το Ιράκ, θα το δούμε αυτό. Δεν είναι καθόλου μικρή χώρα, άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν θέλουμε να δουλέψουμε στη Βαγδάτη και να είμαστε πιο παρόντες και να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα ε, ως προς το έργο μας, θα χρειαστούμε περισσότερους πόρους. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν καταβάλει προσπάθεια σε σχέση με τις συστάσεις που προέκυψαν από την στρατηγική αναθεώρηση. Θα συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και θα δούμε τι θα συμβεί. Μην περιμένετε τίποτα κολοσιαίο να σημειωθεί. Δεν θα γίνει επανάσταση αύριο ε, σε σχέση με τη δράση μας. Δεν θα ε, φέρουμε μια επαναστατική εξέλιξη. Να είστε σίγουροι όμως ότι δεν, κάνουμε εκεί. δεν καθόμαστε εκεί να μην κάνουμε τίποτα. Κάνουμε το μέγιστο που μπορούμε με τους διαθέσιμους πενιχρούς πόρους και με την υφιστάμενη κατάσταση ασφαλείας. Καταφέρνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Με δεδομένο ότι δεν υπήρχε Υπουργείο Εσωτερικών για ένα χρόνο ολόκληρο, που είναι ο βασικός μας ομόλογος, ο βασικός μας εταίρος. Και έχουμε τώρα έναν ε, υπουργό εσωτερικών, ο οποίος έρχεται από την αστυνομία. Οπότε τουλάχιστον θα είναι σε θέση να αντιληφθεί, να καταλάβει τι, τι είναι αυτό που λέμε. Ευχαριστώ. Η ερώτηση μου ήταν διαφορετική. Θεωρείτε κομμάτι των καθηκόντων σας να εντάξετε στην μεταρρύθμιση και τα, τις δυνάμεις ασφαλείας για να μπορέσει η μεταρρύθμιση να, γίνει ένας παράγοντας προσέγγισης των ΣΥΙΤΟΝ και των Σουνιτών. εντάσσοντας δηλαδή τις δύο ε, θρησκευτικέ αυτές ομάδες στην ε, αστυνομία. Δηλαδή δεχόμαστε το ότι το Υπουργείο θέλει να χτίσει μια αστυνομία που θα βασίζεται αποκλειστικά στους ΣΥΙΤΕΣ. Δεν έχω τέτοιο ε, τέτοια εικόνα. το κατά πόσον η, στην, ε- κατά πόσον ε, παράγοντας ενότητας και ε, ενίσχυσης της αστυνομίας είναι μια ενιαία αστυνομία είναι προφανές πως ναι. Δεν μπορούμε όμως να το επιβάλλουμε από πάνω. Το να προσπαθήσουμε μαζί με τις τοπικές αρχές εντός και εκτός της βαχδάτης συζητώντας τα, τα, τα ίδια επιχειρησιακά, όχι πολιτικά θέματα, να βρούμε κοινή, κοινές λύσεις μεταξύ των διαφόρων πλευρών για να χτίσουμε μια κοινότητα αστυνομίας που σε 10, 20, 30, 40, δύο ίσως χρόνια αν είμαστε τυχεροί να λειτουργήσουν ενωτικά η απάντηση μου είναι ναι. Μπορούμε. Θέλει όμως μεγαλύτερη εμπλοκή. Εγώ σας είπα έχω ε, μια εμπειρία από τη Βοσνία. Διαφορετικά ήταν η κατάσταση εκεί, αλλά εν τέλει είχε τρει εθνοτικέ ομάδες και 15 αστυνομίε. Δεν λέω ότι η κατάσταση στο Ιράκ ήταν χειρότερη από ό,τι στην Βοσνία. Αλλιώ βέβαια η κατάσταση της ασφάλεια στην Βοσνία. Οι αλλαγέ όμω που κάναμε ήταν με μία προσέγγιση όχι από... Ξεκινήσαμε από πάνω προς ε, τα κάτω, δεν πετύχαμε τίποτα και μετά αλλάξαμε από κάτω προς τα πάνω. Με καλά, όχι τρελά, αλλά καλά αποτελέσματα. Το να δοκιμάσουμε το ίδιο σε μια χώρα όπως το Ιράκ δεν ξέρω αν θα πιάσει, αλλά μπορεί να το δοκιμάσουμε. Κύριε Νόημαν. Ευχαριστώ. Μία δική μου ερώτηση δεν απαντήθηκε. Αφορούσε το διάλογο με τους διαδηλωτές. Δεν είναι στην εντολή σας. Έχετε όμως στενές σχέσεις με την αντιπροσωπεία της Ένωσης και επηρεάζει τη δουλειά του Υπουργείου αν θα έχουμε για μήνες ε, καταστολή διαδηλώσεων με δακρυγόνα κλπ. Τι άποψη έχετε όπως είπα και στην πρώτη μου εισήγηση, η Ένωση έχει μία σχέση με την κοινωνία των πολιτών που ενισχύεται. Μέσω του διαλόγου θα φτάσουμε και σε άλλους παράγοντες για ζητήματα ασφάλειας. Τώρα, να προσεγγίσουμε τις διαδηλωτές, απαντώ όχι. Θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για μας. το να περνάμε μηνύματα ή να παίρνουμε μηνύματα από τους διαδηλωτέ είναι άλλο θέμα. Η κατάσταση ασφαλείας αυτή τη στιγμή μας περιορίζει κάπως. Αλλά η κατάσταση βελτιώνει σταθεροποιείται και πιστεύω ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα πάμε προς μια μεγαλύτερη παρουσία μας επιτόπου, κάτι που θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας να προσεγγίσουμε και άλλες πλευρές. Ευχαριστώ πολύ τους δύο ομιλητές. Δείξετε, ε, καταλάβετε το ενδιαφέρον της υποεπιτροπής για τα θέματα αυτά. Είμαστε και για την EUEM στο Ιράκ και γενικότερα για την κατάσταση στο Ιράκ και την παρουσία των διαφόρων ευρωπαϊκών, των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Σας ευχαριστώ για τις ε, απαντήσεις Ξέρω ότι είστε υποχρεωμένοι να εκφράζεστε μόνο για τις δικές σας αρμοδιότητες. Αλλά υπάρχουν δεσμεύσεις και δεσμεύσεις. Τραβήξτε το όσο μπορείτε. Σας ευχαριστώ εκ νέου. Chers collègues, je Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην εξή αρχή. Όσοι καθυστερούν δεν θα πρέπει να τιμωρεί η καθυστέρησή τους σε αυτούς που είναι ήδη παρόντες. Ε, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση από μια ομιλήτρια, η οποία όμως μας έχει ενημερώσει και άρα μπορούμε ήδη να ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με τα 10 χρόνια της PSDC, της... Ε, γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε μαζί μας τον Κρίστεφε Μέγερ, καθηγητή για αρμόδια θέματα, σχετικά θέματα στο King's College του Λονδίνου, που θα μας ε, μιλήσει για αυτό το θέμα. Έχουμε τον πρέσβη Πιέχ Βημό, πρώην πρέσβη της Γαλλίας, ε, πρώην Γενικό Γραμματέα του SAE, και ε, senior εφηγητή στο Ίδρυμα Carnegie στο ε, τμήμα για την Ευρώπη και έχουμε και τον κύριο Μπρουκ Στίγνερ, δημοσιογράφο και αναλυτή στο James Defense Weekly. Ο καθηγητής Μέγερ θα μας παρουσιάσει τέσσερις σύντομες μελέτες έτσι όπως το ζητήσαμε και θα μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις για τις πρόσφατες εξελίξεις για θέματα ασφάλειας και άμυνας κοινή πολιτικής αυτών και θα μας μιλήσει για τις μελλοντικέ προοπτικές. Έχετε λάβει όλοι σας αυτές τις μελέτες αν δεν απατώμε. Θα μας τις παρουσιάσει και θα αποτελέσει αυτό αντικείμενο για ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων για τις επιχειρήσεις, για τη ε, δυνατότητά μας στην αμαντική, για την βιομηχανία, για το θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα ευρύτερα. Προτείνω λοιπόν να του δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο, να πάρει το λόγο πρώτος ο κύριος Κρίστοφερ Μέγερ και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους βουλευτές που ενδιαφέρονται να του θέσουν ε, ερωτήματα και μετά θα έχει έρθει η Ναταλή Τοτσί ενδεχομένω θα πάρει το λόγο και θα ακούσουμε και τον κύριο Τίγνερ και μετά θα ακούσουμε του βουλευτέ που θέλουν να του θέσουν ερωτήματα. Κύριε Μέγερ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τη δουλειά μας. Πρόκληση είναι για μένα να παρουσιάσω σε 15 λεπτά 45 σελίδες ενημερωτικών σημειωμάτων για θέματα πολιτικής. Έχω και τον συνάδελφο κύριο Τζόνς που είναι εκεί στο βάθος της αίθουσας, ο και Μπεν Βίλκινς και Σοφία Μπάσεφ είναι εδώ οι συνεργάτες ε, θα συμπληρώσουν αν ξεχάσω κάτι. Βεβαίως πρέπει να λειτουργήσω επιλεκτικά, ε, να διαλέξω και να μιλήσω για τα, τους τις πιο έντονες προκλήσεις, τους πιο ε, σημαντικούς τομείς πολιτικής. Ελπίζω να είναι η συζήτηση παραγωγική. Και εκφύσεως βεβαίως θα αναδείξω τα προβλήματα και δεν θα επενέσω τα επιτεύγματα ε, για τα δέκα χρόνια της ε, πολιτικής αυτής. Σίγουρα η πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα έχει ε, διανύσει μεγάλη διαδρομή, ειδικά αν δει κανεί ε, τα πρώτα χρόνια 2003-2006, έτη κατά την οποία έγιναν οι πρώτε στρατιωτικέ επιχειρήσει. Ε, στην αρχή η συνθήκη τη Λισαβόνα φάνηκε να καθυστερεί την ορμή που δόθηκε στην κοινή αμυντική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Τώρα όμως έχει υπάρξει νέα ορμή. Νομίζω και ελπίζω ότι αυτά τα ενημερωτικά σημειώματα βοηθούν να λειτουργεί κανείς ρεαλιστικά, να έχει ένα σωστό προβληματισμό στις σωστές βάσεις και να βλέπει τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες της κερδής πολιτικής. Και ελπίζω ότι οι σκέψεις μας θα βοηθήσουν για να, ε, έτσι ώστε οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται να οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις ε, που να λειτουργούν και να μην υπάρξει μόνο μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω αποκομμένη από την πραγματικότητα του εδάφους. Μιλούμε για τις ε, επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας αλλά και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το πολιτικό σκέλος των επιχειρήσεών μας έχει, έχει πετύχει τους περισσότερους στόχους του. Απλά οι στόχοι αυτοί δεν, δεν ήταν πολύ ευρύ. Ε, για παράδειγμα, στη Σομαλία ε, δείχνουμε είδαμε και δείξαμε πώς μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική, να πετυχαίνει διάφορους στόχους ε, ταυτόχρονα. Τον ανθρωπιστικό στόχο, προστασία των τροφίμων ε, που έρχονταν με τα σκάφη, τον, ε, τα αντίστοιχα, διατήρηση των εμπορικών θαλάσσιων διάβλων επικοινωνίας ανοιχτών, διατηρήση ανοιχτών αυτών των διάβλων, αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της πειρατείας, ε, των αδύναμων κρατών και της αστάθειας, ε, φαινόμενα που επικρατούσαν στο, κέρος, στο κέρας της Αφρικής. Αυτή ήταν, αυτή ήταν η στόχη μας στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας και τους πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό στη Σομαλία. Βλέπετε το παράδειγμα επιτυχημένο. Και σίγουρα... Ε, φαίνεται ότι είναι πολύ προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δρά, αλλά φαίνεται να μην υπάρχει πολιτική βούληση να το κάνει. Το είδαμε αυτό στη Λιβύη το 2011 και στο Κονγκό το 2012, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν έτοιμη και δεν ήθελε να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να μην χρησιμοποιήσει τα τάγματα, ε, τα στρατιωτικά που διέθετε. Χρειάζεται χρόνο από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση μέχρι ότου να δημιουργηθούν οι πόροι που θα οδηγήσουν στη στήριξη της εφαρμογής τη απόφαση αυτή. Χρειάζεται χρόνος ε, εν τω μεταξύ να απαντηθούν αυτά στις αντίστοιχες διασκέψεις και άπαξ και απαντηθούν και ρυθμιστούν να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι επί Το 80% των πόρων ε, έχουν επιτευχθεί για το σύνολο των πολιτικών. Κατά μέσο όρο το 30% είναι αυτό που συμβαίνει κανονικά. Ορισμένες λύσεις για να Υποτίθεται ότι θα πρέπει το 80% μπορώ να καλύπτονται, αλλά τελικά το 30% φτάνουμε να καλύπτουμε και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και τη λειτουργία ε, πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα χρηματοδότησης. Αυτό σίγουρα ισχύει. Κάτε με ε, Ένα τομέα στον οποίο είναι απαραίτητο να σημειωθεί πρόοδος είναι η καλλιέργεια στρατηγικής κουλτούρας και νοοτροπίας στο στρατιωτικό τομέα, όπου οι ευρωπαϊκές αποστολές ήταν πολύ λιγότερο πολυάριθμες από ό,τι οι πολιτικές αποστολές πολιτικής προστασίας. Πολύ περισσότερα δηλαδή πρέπει να γίνουν για να υπάρξει σύγκληση της χρήσης αυτών των μέσων για να αντιμετωπιστούν οι απειλές στην ασφάλεια ε, σύγκληση ευρωπαϊκή να έχουμε μια κοινή αξιολόγηση, αυτό θα είναι καθοριστικό. Άρα οι υπηρεσίε πληροφοριών είναι ακρογωνίες λίθος για ε, το να μοιραζόμαστε πληροφορίες προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την απειλή. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι να αξιοποιήσει καλύτερα τους υφιστάμενους πόρους, γιατί οι αντιπροσωπείες δεν αξιοποιούνται με το βέλτιστο δυνατό ε, τρόπο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το μοίρασμα δηλαδή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Ίσως να, ίσως να ακολουθήσουμε τη νομική οδό της ενισχυμένης συνεργασίας δηλαδή με μικρότερο αριθμό κρατών μελών, οι οποίες, τα οποίες μέλη να θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών και της ανταλλαγής των πληροφοριών αυτών. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας έδωσε νέες ευκαιρίες και η πολιτική, εξωτερική πολιτική ασφάλειας και συνεργασίας και το ΠΕΣΚΟ, ε, δηλαδή τα κοινά συμβούλια όπως γνωρίζετε, ήταν κάτι το πολύ σημαντικό. Έχουμε ε, το υπερεθνικό και το διακυβερνητικό σκέλος και η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αποτελεί πρόβλημα για το θεσμικό πλαίσιο. Πολλές ε, λύσεις μπορούν να δοθούν σε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να επινοήσουμε πιο ευέλικτες αλλά συνδεδεμένες μορφές διαδικασίας λήψης αποφάσεων με μικρότερο αριθμό κρατών μελών και όχι με το σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και μέρος άλλωστε του ΠΕΣΚΟ ε, και ε, είναι και μέρος της πρωτοβουλίας για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, όποια μορφή και αν πάρει αυτό. Ένα από τα ωφέλη ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας θα ήταν το εξής. Ε, θα έπρεπε να είναι μια πιο άτυπη μορφή και να συνεχίσει να έχει δεσμούς και με το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά το Brexit. Μετά μπορεί να επικταθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία ε, σε ορισμένους κλάδους. Μιλούσαμε για τις κυρώσεις ή για τις αποστολές πολιτικού και όχι στρατιωτικού χαρακτήρα. Εκεί θα μπορούσαν να αποφασίζονται αυτές όχι με μονοφωνία αλλά με ειδική πλειοψηφία. Και να έχουμε και τη ε, και ε, ρήτρα που θα δίνει τη δυνατότητα να αναλάβει κανείς περαιτέρω δράση από μόνος του, άπαξ υπάρχει ομοφωνία για τον ευρύτερο στόχο είναι, πρέπει να είναι πιο ταχύρυθμη η διαδικασία λύση των αποφάσεων για να φαίνεται η βούληση ανάληψης δράση και να μην υπονομεύεται η στήριξη και η επίκληση στην αλληλεγγύη και, αλλά να μην υπονομεύεται και η θεσμική οντότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, στην περίπτωση κατά την οποία λιγότερα κράτη-μέλη θα θελήσουν να κινηθούν πιο ομαδικά και πιο ξεχωριστά για να προχωρήσουν περισσότερο από τα υπόλοιπα. Τώρα, ως προς τις δυνατότητες Παρά την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική και παρά το σχέδιο το εφαρμοστικό για τα της αμήνης ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχουν δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι σημαίνει αυτό για τις προτεραιότητες των κρατών μελών ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αν διαβάσει κανείς την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Συνολική Στρατηγική βλέπει ότι η στόχη είναι πολύ πιο φιλόδοξη από ε, το, το στόχο του Πίτερσμπεργκ. Δεν είναι σαφές όμως τι προσδοκά πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει να έχει στρατηγική αυτονομία από τις Ηνωμένες Πολιτείες 100% γιατί αν επιθυμεί να πετύχει κάτι τέτοιο οι επιπτώσεις είναι δραστικές και πολύ σημαντικές αν θέλουμε να σημειώσουμε μεγάλη προόδο, σίγουρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερο, να δαπανίσουμε περισσότερα και πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα το θέμα του εξορθολογισμού. Ε, αμυντική συνεργασία σε, αμοιβαίο, σε αμοιβαία βάση μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις ε, επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Ε, βοηθάει και αυτό που μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολύ χρήσιμο, να καλύψουμε το κενό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Παγκόσμιας Στρατηγικής και μιας λευκής βίβλου ευρωπαϊκής για θέματα αμήνης, όπου θα παριθμούνται τα θέματα πολύ πιο περιστατωμένα, πολύ πιο λεπτομερή. Ορισμένα κράτη-μέλη μίλησαν για το ενδεχόμενο ύπαρξη στρατηγικής εξίδας. Τι θα, θα μπορούσε όλο αυτό να περιλάβει, τέλος πάντων. Ε, τώρα, για τα θέματα των δαπανών, σύγκριση γίνεται πάντα με τα νούμερα των Αμερικανών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλότερο επίπεδο δαπανών οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όμως, μήπως υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Η, 20 έχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 20 καταδρομικά, η Αμερικανοί 6, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 16 πολεμικά ε, πλοία υψηλών δυνατοτήτων, η Αμερικανοί μόνο 3 και το καθεξής. Ε, η οικονομία κλίμακας είναι σημαντική. Πρέπει να έχουμε οικονομία κλίματος, πρέπει να στηρίξουμε τη διαλειτουργικότητα και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση. Το EDF είναι ένα νέο σημείο κίνησης για να ενισχύσουμε αυτές τις δεξιότητες και να χτίσουμε ε, αυτή την αμυντική αγορά θα φτάσουν οι σημερινές δαπάνες για να μετατρέψουμε το τοπίο, να αλλάξουμε το σκηνικό. Νομίζω ότι απαντάτε αυτό στο κείμενό μας. Παραμένει όμως η πρόκληση. Αν θέλουμε να φτιάξουμε την EDTIB, τότε πρέπει να αλλάξει ριζικά η ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, αλλά και η αμυντική πολιτική του κάθε κράτους μέλους. Πρέπει να δούμε το θέμα των εθνικών προτιμήσεων στις κρατικές προμήθειες στρατιωτικού υλικού. Να αναθεωρήσει κανείς. Το 80% των αμυντικών δαπανών παραμένει εθνικό, ε, σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι τεράστια πρόκληση. Επομένως, και το τελευταίο που θα ήθελα να πω έχει να κάνει με την πρόσβαση τρίτων μερών στο EDF το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και κατά πόσο μπορούν να συμμετάσχουν και αμερικανικές ή αγγλικές ε, αμυντικές εταιρείες. Άλλο μεγάλο πρόβλημα για την ανάληψη πρωτοβουλειών στο τομέα αυτό. Άρα, συμπερασματικά, τι λέει το ενημερωτικό μας σημείωμα. Πρέπει να κάνουμε πιο αποτελεσματική την πολιτική μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις φιλοδοξίες που, με τις οποίες έχει επιφορτιστεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για να γίνουν αυτά θα χρειαστεί χρόνος, θα χρειαστεί αλλαγή νοοτροπίας σε διάφορα επίπεδα και θα χρειαστεί ε, ε, περισσότερη σύγκληση μεταξύ εθνικών αρχών. Ε, θα πρέπει οι εθνικοί εταίροι να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό των Βρυξελών. Όμω, αυτή η στόχη είναι μακροπρόθεσμη. Προκλήσει θα έχουμε και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Όταν συνέταξα την έκθεσή μου για την αναθεώρηση των επιχειρήσεων με βάση αυτή τη πολιτική, αναρωτήθηκα, ερχόμαστε μήπως να λύσουμε τα προβλήματα των χθεσινών επιχειρήσεων που οργανώσαμε, οι οποίες όμως έχουν λήξει πλέον. Μήπως δεν έχουμε αντιληφθεί τα αυριανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που θα συγκροτήσουμε για μεθαύριο. Δεν είχαμε τρομακτική αποτυχία. Εάν όμως είχαμε ένα μογκα ένα σενάριο τύπου Μογκαντήσου ή τύπου Σρεμπρένιτσα ή τύπου Φαλούτζα, δηλαδή γεγονότα στα οποία, τα οποία συνέβησαν πριν να έχουμε κοινή αμυντική πολιτική. Ε, θα ήμασταν σε θέση να λειτουργήσουμε, να αντιδράσουμε να είναι έτοιμη η ευρωπαϊκή πολιτική να παρέμβει, υπάρχει πολιτική βούληση, έχει τις δυνατότητες να δράσει αν έχουμε ξέσπασμα τέτοιων ε, σενάριων απειλητικών. Έχουμε νέες προκλήσεις, νέες απειλές και πρέπει να τις γνωρίζουμε. Στο παρελθόν ε, ήμασταν πολύ υπεραισιόδοξοι και σε θέματα αμυντικά και σε άλλους τομείς πολιτικής. Το να είναι κανείς προνοητικός σε στρατηγικό επίπεδο είναι βασικό για να έχει επιτυχημένη άμυνα τα επόμενα δέκα χρόνια. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων λοιπόν. Η πράσινη χαρανόημα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω που μπορεί να αναφέρεται όμως και στους άλλους ομιλητές. Υπήρξε μεγάλη μείωση της, του σύνθετου χαρακτήρα των ε, αποστολών ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Η Άρτεμις, η αποστολή στην Μακεδονία ε, δεν υπάρχουν πια, ενώ αυξάνεται η βία και η ένταση στη γειτονιά μας. Από την άλλη όλοι λένε ότι πρέπει να απαντάμε σε όλες τις συγκρούσεις, να, γίνονται, να, να υπάρχει παρέμβαση και δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί δεν γίνονται. Μιλήσατε για Φαλούτζα, Σεμπρένιτσα. Έχουμε το Ιντλιμπ Παρόμοιες περιπτώσεις γενοκτονίας έχουμε, απλώς τις αγνοούμε. Ο κύριος Γκάλ για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ και θα μιλήσω γερμανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισκόπηση αυτή που μας δώσατε. Και συμφωνώ γενικά με την παρουσίαση που κάνετε. Εγώ έχω δει ότι από την θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνα όντως τα πρώτα πέντε χρόνια δεν ε, ήταν έτσι, αλλά μας βοήθησε ο Βλάντιμιρ. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν ε, ένα, μια αφορμή όπου διαπιστώσαμε ότι και στην άμεση γειτονία μας μπορούν να συμβούν πράγματα τα οποία έχουν ε, εμέσως επιδρασή και σε εμάς. να κάνω μία παρατηρήση για κάποιες ε, πτυχές που αναφέρατε. Intelligence sharing, μυστικές πληροφορίες. Θεωρώ ότι αυτό δεν μπορεί να μπει σε μια τυποποιημένη διαδικασία. Μιλήσατε για ενισχυμένη συνεργασία. Νομίζω ότι όντω μόνο εθελούσιο μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα στι Βρυξέλλε, όντω. Όπου και να λαμβάνει χώρα αυτή, θα πρέπει να υπάρχει ένα μέρο όπου όλοι θα ξέρουν ότι αν κλείσει μια συνάντηση, μπορούν να έρθουν όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και που θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σκόπιμο ως λύση. Πιστεύω ότι όντω θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τις πλειοψηφικέ αποφάσεις. Είτε μιλάμε, ε, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις κυρώσεις, αν κατά πόσο έχει νόημα η συζήτηση αυτή. Εντάξει, αν φτάσουμε μέσω εκεί βλέπουμε. Συμφωνώ. Μια άλλη λύση θα ήταν να υπάρξει μια επικοδομητική αποχή. Να πούμε δηλαδή ότι κοιτάξτε θα ακολουθήσουμε την ε, οδό τη αποχή, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε, αλλά θα αφήσουμε τους άλλους να προχωρήσουν. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του δύο πόρου ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξία. Το επίπεδο φιλοδοξία ε, θα πρέπει να προσανατολιστεί την ε, ανάλυση του επίπεδου ασφάλειας για να δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις σε ό,τι αφορά τις ε, δυνατότητες θα πρέπει να έχουμε δυνατότητες ε, πλήρους φάσματος, full spectrum. Μιλήσατε για στρατηγική αυτονομία τώρα, κυρίως στο ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε όμως μαζί μου ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Λιβύη αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα, όπου θα έπρεπε να το παίξουμε στα σίγουρα. Για να κάνουμε κάτι στη Λιβύη, να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του ΝΑΤΟ, ένα απλό βέτο του Ερντογάν θα αρκούσε για να τα θέσει όλα στον πάγο. Θα μπορούσαμε λοιπόν ο Ερντογάν να, μπλοκάρει τα πάντα με ένα ενδεχόμενο βέτο και από πλευρά στρατηγικής αυτονομίας ε, αυτή είναι η προορισμή. Αυτά. Ίσως ξέχασα και κάποιες ερωτήσεις, αλλά ενδεχομένω στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος. Ο κύριος Βασέσκου. Θα Συνεχίζω σε αυτά που είπε ο κ. Γκέλερ. Είναι ασαφέστατο, κατά την άποψή μου, τι θα πει στρατηγική αυτονομία. Εγώ είμαι παλιός πρώην αρχηγός κράτους, μέλους του ΝΑΤΟ, μέλους της ΕΕ. Οι δυνάμεις μας ήταν πάντα στη διάθεση του ΝΑΤΟ. Δεν δημιουργήσαμε ποτέ στρατιωτικούς πόρους που θα ήταν στη διάθεση της Ένωσης. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι οι περισσότερες από τις 22 χώρες της Ένωσης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ έχουν την ίδια προσέγγιση. Υπό τους όρους αυτούς πόσο αυτόνομοι μπορεί να είμαστε όταν τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Διότι αν παίζουμε με τους πόρους, σε κάποια στιγμή μπορούμε πρώτον να απονομιμοποιήσουμε το ΝΑΤΟ, αφαιρώντας ε, τις ε, δυνάμεις από το προγραμματισμό του ΝΑΤΟ. Αυτή την έννοια κάποια στιγμή πρέπει να την ε, διευκρινίσουμε. Από την άλλη πλευρά βέβαια συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να εισαχθεί η αρχή της πλειοψηφίας της αποφάσεις. Αλλιώς θα μείνουμε, εγώ έχω εμπειρία από τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, δύο-τρεις χώρες μπλόκαραν αποφάσεις σημαντικές αποφάσεις. Πρέπει να εισάγουμε τον κανόνα της πλειοψηφία. Όταν δεν βλέπουμε τη στρατηγική πραγματικότητα αυτές τις μέρες, ίσως να μπορούμε να αναπτύξουμε χωριστούς πόρους έτοιμους για ευρωπαϊκή παρέμβαση. Αλλιώς, αν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας στη σωστή στιγμή, η σημασία μας θα μειώνεται συνεχώς. Δεν είναι αρκετό να είμαστε ηγέτες τα οικονομικά. Είναι σαφές ότι αυτό το καιρό οι μεγάλοι παίκτες έχουν Οικονομία και στρατό. Ευχαριστώ. Ο Κρίς Πέτρας. Ε, ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μία συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Συμφωνώ όμως ότι όταν τα συμφέροντα της Ένωσης και του ΝΑΤΟ, της Ένωσης και των ΙΠΑ δεν συμπίπτουν, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα αυτόνομης δράσης. Αυτό στο μέλλον θα γίνει συχνότερο από ό,τι τώρα. Και συμφωνώ με όλα τα σημεία που αναφέρατε. Για μένα όμως η πρώτη ερώτηση είναι όταν η πρόεδρος της Επιτροπής είπε χρειάζομαι μια γεωπολιτική επιτροπή και αυτή η επιτροπή θα είναι γεωπολιτική, το ερώτημα είναι τι σημαίνει. Ποιο είναι το όραμα του Συμβουλίου, της Επιτροπής, τέλος πάντων να είναι, για το τι σημαίνει γεωπολιτική εικόνα του κόσμου. Πότε, πότε παρεμβαίνουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η γεωπολιτική εικόνα που έχουμε για το μέλλον και τι θα κάνουμε για το μέλλον. Χρειάζεται μεγαλύτερο περιεχόμενο η δήλωσή μας ότι είμαστε γεωπολιτικοί. Ξέρετε, θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε, αλλά ξέρετε, θα ήταν ακόμα πιο ε, προβληματική θα σαν είσαι σαν γιατί θα έπρεπε να σε 1,5 λεπτό να σχολιάσετε μία έκθεση για τα 10 χρόνια της ΕΠΑ. Θα δώσω το λόγο σε, στους άλλους ομιλητές ζητώντας τους όχι μόνο να παρέμβουν αλλά και να μας πούν τα, την άποψή τους για αυτά που ήδη ακούστηκαν. Ο κύριος Γκάλερ θα έξανα το λόγο. Μην ξεχάσετε να θέσετε και την ερώτηση όμως. Θα το δώσω μετά. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Ο Μπεν Τζόνς ε, νομίζω θα απαντήσει στην ερώτηση του κύριου Μπασέσκου για τη στρατηγική αυτονομία, αν το επιτρέπετε πρόεδρε. Τι έγινε με γιατί δεν είναι τόσο σύνθετες οι αποστολές ΕΠΑ. Πολλά πράγματα έγιναν. Πρώτον, η Ένωση πολιτικά αποπροσανατολίστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των αμυντικών δαπανών. Υπήρχε δηλαδή ένα οικονομικό πρόβλημα και ένα πολιτικό πρόβλημα, έλλειψη ηγεσία ενδεχομένω στο θέμα των αποστολών. ΕΠΑ. Η εμπειρία της Λιβύης ήταν απογοητευτική για κάποιους. Η γερμανική εμπειρία σκοτίνιασε λίγο τον ενθουσιασμό των ΕΠΑ. Ίσως η κρίση που αντιμετωπίζει η Ένωση στα σύνορά της είναι τόσο έντονη που η Ένωση έχει επιφυλάξεις στον έμπλακη. Αν θέλουμε να είμαστε γεωπολιτικοί στη Λιβύη και τη Συρία, ή εναντί της Ρωσίας μπαίνουμε σε μία πρόκληση που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να ανταποκριτούμε. Υπάρχει πάντως ε, τώρα μία ετοιμότητα να προχωρήσουμε. Αυτό το δείχνει και η συζήτηση για τη Λιβύα. Τώρα για την ε, αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Ενισχυμένη συνεργασία δεν σημαίνει ε, υποχρεωτική, αλλά εθελούσια ανταλλαγή πληροφοριών. Απλώς θα δίνει μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των κρατών μελών και χρειάζονται νέα κράτη-μέλη. Δεν φεύγουμε δηλαδή από την αρχή της εθελούσιας ανταλλαγής ε, πληροφοριών, απλώς υποστηρίζουμε την σωστή υποδομή γι' αυτό. Να δώσω το λόγο στον Μπέναν αν γίνεται για, την στρατηγική, για τη στρατηγική αυτονομία. Ναι κύριε Τζόνς, ε, μα θέλετε... Μου δίνετε τις εύκολες ερωτήσεις. Καταρχάς, τι εννοούμε με τον όρο στρατηγική. Κανείς δεν νομίζει να προτείνει η Ένωση να αναπτύξει τις ικανότητες της, ικανότητες σε δύο βαθμό που είναι πλήρως αυτόνομη στην άμυνά της. Δεν νομίζω ότι προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι σημαίνει στρατηγική αυτονομία. Ένα παράδειγμα αυτόνομης δράσης ήταν από τη ΣΥΠΑ στην Λιβύη που ξεκίνησε από Γαλλία ε, Βρετανία και αυτή η επιχείρηση δύσκολα, πολύ δύσκολα θα είχε ολοκληρωθεί από τις δύο αυτές χώρες αν δεν είχαν παρέμβει και συμβάλει είπα. Άρα η αυτονομία σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε περιπτώσεις όπως την εξαρτία στη Λιβύη μια άλλη επιχείρηση που θα μας επιτρέπει να ορίσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Γιατί ο όρος στρατηγικό σημαίνει πολλά πράγματα σε πολλούς. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω και την Αταλή Τότσι. Ας περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της συζήτησης αυτής. Ο Πιέρ Βημό έχει, έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και δεν θα ήθελα να σας απασχολήσω. Πολύ ώρα, Γιατί έχουμε και πολλούς άλλους ομιλητές που θα ήθελα να πάρουν το λόγο και προφανώ έχουμε και πολλέ ερωτήσεις, οι οποίε θα πρέπει να απαντηθούν. Να, αναφερθώ όμως σε αυτά που μόλις ακούσαμε. Για το πόσο περίπλοκο είναι το θέμα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα τόσο περίπλοκα που σε ένα βαθμό έχουμε την εντύπωση και εγώ προσωπικά έχω την εντύπωση ότι έχουμε όλο και πιο πολλά εργαλεία, όλο και πιο πολλέ ιδέε, όλο και πιο πολλά ε, δομές συνεργασίας στα, πλαίσια τη πολιτική ασφάλεια και άμυνα. και εκ παραλλήλου κάποιε από τι πιο μεγάλε κρίσει που αντιμετωπίζουμε βρίσκουν την Ευρώπη σε μεγάλη δυσκολία δεν ε, μπορεί να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή σήμερα. Κοιτώντας αυτά που γίνονται σήμερα στον Περσικό κόλπο, στη Λεβύη, στη Σαχέλ, όλο και πιο πολύ αναφέρουμε το πόσο απαραίτητο είναι να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε ότι οι Υπουργοί Άμυνας, οι Υπουργοί Ιστορικών προσπαθούν να κινητοποιηθούν και εκ παραλλήλου διαβλέπουμε και μία, ένα δισταγμό, μία προθυμία μεταξύ των κρατών ε, μελών. Κάποιοι έχουν πιο πολύ ενέργεια από ό,τι άλλους και γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε. όπου σε κάποιο βαθμό δεν μπορούμε να συνδέσουμε όλα τα διαφορετικά στοιχεία που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε την ε, παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε πώς συγκεντρώθηκε ξαφνικά μια νέα ορμή για την ε, ΚΕΠΑ. Το 2013 ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την πολιτική άμυνας και ναι, εξωτερική πολιτική πήρε πέντε λεπτά όλη και όλη η συζήτηση. Είχαν προφανώ και πολλά άλλα να συζητήσουν. Μπήκε στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν έδωσε κανένα ιδιαίτερη σημασία. Και σήμερα, όπω είπατε και εσεί, έλαβε χώρα η κρίση στην Ουκρανία. Έγινε το δημοψήφισμα για τον Brexit, οι Αμερικανικές εκλογές και εντελώς ξαφνικά όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώθηκαν στην πολιτική Ασφάλεια και άμυνας, το EDF, το PESCO και πολλά άλλα στοιχεία. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ειρήνη. Και παρά όλα αυτά, εξακολουθούμε να έχουμε την εντύπωση ότι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατεπίγουσα κρίση και χρειάζεται να δώσουμε ε, άμεσα απαντήσεις στις ε, προκλήσεις της εκάστοτε, βρισκόμαστε πάλι εκεί που ήμασταν πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Και άρα αυτό που θέλω να θέσω είναι το εξή. Αντιμετωπίζουμε πολλά μεγάλα ζητήματα και δεν ξέρουμε τι απάντηση να δώσουμε στην παρούσα φάση. Καταρχά για θέματα κυριαρχία. Τα πολύ χρήσιμα έγγραφα τα οποία μας παρουσίασε ο καθηγητής Μέιορ έχουν να κάνουν με αυτό. Κατά πόσον θέλουν να διατηρήσουν κυριαρχία τα κράτη-μέλη σε τα θέματα αυτά ή κατά πόσον προτίθενται να μοιραστούν την κυριαρχία αυτή με άλλους. Εδώ φυσικά τα όρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια λύση. Και να πω ότι πολλές από τις κρίσεις που διανύουμε σήμερα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Βλέπουμε μια πάρα πολύ ευέλικτη πολιτική ασφάλειας και αμα άμυνα. Βλέπουμε στην αυτολία και στον Περσικό κόλπο. Στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του οποίου προέδρευσε η Φραγκελίκα Μογκερίνη, υπήρξε αυτή η ιδέα να μετακινηθούν τα κράτη-μέλη και να διαδραματίσουν τον ρόλο ηγετικών κρατών ε, στα ναυτιλιακά με αμοιβαία χρήση πληροφοριών και με κοινή ευθύνη. Είχαμε τη Γαλλική Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία παρέμβαση, ονομάζεται. Έχουμε τις επιχειρήσεις στο ΣΟΧΕΛ όπου οι χώρες που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις καλούνται να συμμετέχουν και έτσι πέρα από τις 28 από την Βαύρη 27 κρατών μελών θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της πραγματικότητας της εκχώρησης κυριαρχίας το οποίο δεν είμαστε σε θέση να το επιλύσουμε με απλό τρόπο. Κατανοητό. Δεύτερο θέμα, η ταυτότητα. Και εδώ δερχόμαστε κρίση. Τι θέλουμε να κάνουμε με αυτή την ε, νέα αρμοδιότητα στην πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Είναι εντυπωσιακό, κοιτώντα ε, τα καθήκοντα του Πίτερσμπουργκ και αυτά που περιλαμβάνονται στην συνθήκη της Λισαβόνας, έχετε τα θέματα ειρήνευσης και διατήρησης της ειρήνης και βλέπουμε πόσο σταδιακά και με πολλή υπομονή υπησέρχονται και άλλα καθήκοντα που έχουν να κάνουν με στρατιωτική καθοδήγηση και παροχή συμβουλών, ανθρωπιστική α, βοήθεια κτλ. κτλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι θέλουμε να προχωρήσουμε να προχωρήσουμε πραγματικά. Στο σημείο αυτό αρχίζουν να κάνουν πίσω και να διστάζουν τα κράτη-μέλη και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό τελικά είναι πραγματικά ευθύνη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ λοιπόν αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Κατά τρίτον, έχουμε μια πολιτική και στρατιωτική στρατηγική. Αυτό που ήταν σαφέ στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική στην παγκόσμια στρατηγική ήταν ότι επιμένουμε σε, στο σκέλος της ασφάλειας και της άμυνας και όλα τα στοιχεία αυτά που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται μέσα από τα διάφορα εργαλεία και τα διάφορα μέσα τα οποία εφήβραμε, ε, είχαν μία έλλειψη. Μία σαφής απάντηση σε κάποια ξεκάθαρα ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις ε, επιχειρήσεις αυτές τις οποίες θα μπορούσα να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δράσει πραγματικά ως παγκόσμιος παράγοντας. Ε, επανερχόμεθα στο θέμα της στρατηγικής αυτονομίας κρίσης, όπου ούτε οι Αμερικανοί, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε ο ΟΗΕ είναι σε θέση ή προτίθεντα να παρέμβουν. Και όπου τα ευρωπαϊκά συμφέροντα μα φέρνουν αντιμέτωπου με το ερώτημα ξεκάθαρα κατά πόσον θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει ή όχι. Και πραγματικά αυτό συμβαίνει στην παρούσα φάση. Στον Περσικό κόλπο, στη Λιβύη, στο Σαχέλ, είναι σαφές ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν πολύ ενδιαφέρεται. Ο ΟΗΕ έχει παραδοσιακά το πρόβλημα για είναι αργοκίνητος. Άλλοι φορείς ε, παραμένουν, Τουρκία, Ρωσία και κάποιοι από τους εταίρους και τους φορείς ε, από τον Περσικό κόλπο και η Ευρώπη έχει έντονα την αίσθηση ότι θα πρέπει να είναι παρούσα αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Γιατί δεν έχουμε ορίσει ουσιαστικά τι καθήκοντα προτιθέμεθα να αναλάβουμε σε αυτό το πολιτικό, στρατιωτικό οικοδόμημα. Δεν έχουμε ορίσει το επακριβές επίπεδο φιλοδοξίας που επιθυμούμε. Ακόμα διστάζουμε σε ό,τι αφορά το ρόλο και την ευθύνη που θέλουμε να λάβουμε και κάποια θέματα τέτοια επανειλημμένα οι εταίροι μας, όπως ο ΙΕ, μας έχουν ζητήσει να απαντήσουμε. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ε, συμμετοχή ε, για την οικοδόμηση ειρήνης μαζί με τον ΟΗΕ σε διάφορες περιοχές. Ο ΟΗΕ λοιπόν μας έχει ζητήσει. Μπορείτε να καλύψετε τα κενά από τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει η ανάγκη μέχρι ότου ληφθεί η απόφαση μάλλον από τη στιγμή που έχει ληφθεί η απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ μέχρι ότου καταστεί λειτουργική δύναμη του ΟΗΕ. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει έναν φορέα ο οποίο θα μπορούσε να δώσει απάντηση, αλλά δεν έχουν επιληθεί τέτοια ζητήματα και τέτοιου είδου ζητήματα θα πρέπει να εξετάσουμε. Η Λιβύη λοιπόν αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αν καταφέρουμε να επιβάλλουμε την εκεχηρία και να επικυρωθεί αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ποιο θα είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση και την εποπτεία. εμεί μπορούμε να μεταβούμε επί τόπου ταχύτατα για να τα αναλάβουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει αυτή την υψηλή ευθύνη. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω στο τελική ανάλυση Η μικρή μου παρέμβαση θα καταλήξει λοιπόν στο εξή: Ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χρονική συγκυρία γιατί είναι η στιγμή ανάληψη δράση. Είναι η στιγμή που η Ευρώπη θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσει κατά πόσον επιθυμεί να αποτελέσει γεωπολιτικό παράγοντα ή όχι, όπως το θέσατε και πολλοί από εσάς. Στην παρούσα λοιπόν στιγμή μπορούμε να αποφασίσουμε προς τα πού θέλουμε να οδεύσουμε. Γιατί. Και εδώ θα βάλω τελεία, πρόεδρε, και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ε, ε, τα τελευταία 5-6-7 χρόνια η εντύπωση μου είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική έχουμε παράγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις, έγγραφα επί εγγράφων, χωρίς απαραίτητα μεγάλη σύνδεση μεταξύ τους και χωρίς να ληφθεί τελικά ιδιαίτερη δράση επιτόπου, με εξαίρεση κάποιων πολύ ενδιαφέρουσων ε, ενεργειών και επιχειρήσεων επιτόπου. Αλλά ακόμα δεν έχουμε μπει σε αυτή την πολιτική και στρατηγική στρατηγική που χρειαζόμαστε. Μιλάμε για τη στρατηγική πηξίδα, το πιεσί, Όλα αυτά ξεκινάμε να τα συζητάμε σήμερα. Και υπάρχει... Ε, έχουμε όλε τι αντίξει ότι όλα αυτά θα πάρουν πολύ χρόνο γιατί προφανώ προπετούν και ένα κοινό συντονισμό. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική αυτή ευκαιρία να βλέπουμε μπροστά μας κρίσεις και προκλήσεις που ενδεχομένως να μας αναγκάσουν να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι σκοπεύαμε. Κάποιοι από εσά αναφερθήκατε στο γεγονός ότι η πρώτη ευρωπαϊκή επιχείρηση ήταν πιο εύκολα κατανοητή, μα αυτό ήταν ακριβώς αυτό που είπε και τότε η πατή εκπρόσωπο. να πάμε επί τόπου και να δούμε τι θα κάνουμε. Η Μακεδονία. Η Δημοκρατία του Κονγκό, Αρτεμής και η Αταλάντα Όλες αυτές ήταν επιχειρήσεις όπου προχωρήσαμε χωρίς να κάτσουμε να ρωτηθούμε. Απλά έπρεπε να παραστούμε επί τόπου γιατί μας ετήθηκε και απαντήσαμε σε αυτή την διεθνή έκκληση άμεσα. Θα πρέπει λοιπόν αυτού του είδους την οτροπία, αν θέλετε, να εφαρμόσουμε. Και πιστεύω ότι πραγματικά χρειάζεται πιο έντονα να επικρατήσει αυτή η αντίληψη και αυτή η νοοτροπία. Ευχαριστώ και ζητώ και πάλι συγγνώμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη και να δώσω το λόγο τώρα σε μία από τις ε, βασικές ε, παράγοντες, βασικούς παράγοντες της, ε, της παγκόσμιας της Ευχαριστώ και θα μπορούσα να φύγω, γιατί ουσιαστικά αυτά σκόπευα και εγώ να πω με το προλαλήσατε τα ίδια. Να τα θέσω με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και συμφωνώ. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια διαπιστώσαμε μία μεγαλύτερη δραστηριοποίηση για την ασφάλεια και την άμυνα και μπορούμε να αναφέρουμε μεγάλο κατάλογο με ακρονίμια για πρωτοβουλίες. Έχουν αναλυφθεί, τις ξέρετε όλοι σας και υπάρχουν και κάποιες πρωτοβουλίες εκτό θεσμικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εντό θεσμικού πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημείο εκκίνηση λοιπόν είναι το εξή. Να διαρωτηθούμε γιατί έχουν συμβεί αυτά. Γιατί μετά από μία δεκαετία όπου η πολιτική ασφάλειας και άμυνας είχε χάσει κάπως την ορμή της, είχε χάσει κάπως ε, την έγκλη της, την οποία αναφερθήκατε στο τέλος. Υπήρξε λοιπόν μια στιγμή παρακμής και μετά πάλι πήρε τα πάνω της. Σε τελική ανάλυση νομίζω ότι το θέμα είναι τα εξή τρία. Οι εξή τρει παράγοντε έπαιξαν ρόλο. Καταρχά το θέμα τη ε, ασφάλεια. Ε, Μα ε, καταστράφηκε αυτή η εντύπωση ότι ζούσαμε σε έναν ασφαλή κόσμο Ουκρανία, Συρία, Ιεμένη, Λιβύη. Ήταν σαφή τα αποτελέσματα. Δεν ήταν μόνο το θέμα ότι ήμασταν πιο ανασφαλείς, αλλά είχαμε την αίσθηση ότι ήμασταν πιο ανασφαλείς. Και δεύτερος παράγοντας, ακόμη πιο σημαντικός, ο ρόλος των Ηνωμένων ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Παραμένει ακόμα αντιευκρίνιστος και εδώ το ερωτηματικό ε, είναι όλο και μεγαλύτερο μετά την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά και πριν την εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ ήταν εκεί. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι μιλάμε πραγματικά για ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη ρόλο των ΗΠΑ στο παγκόσμιο προσκήνιο. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ερώτηση. Θα, συνεχίσει, θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να φροντίζουν για την ευρωπαϊκή ασφάλεια τα επόμενα 5, 10, 20, 30 χρόνια. Όπως ξέρουμε όλα αυτά παίρνουν πάρα πολύ χρόνο μέχρι να συσταθούν. Εδώ λοιπόν, έχει, λοιπόν αυτή η ερώτηση. Ακόμα και αν δεν υπάρχει βεβαιότητα και απλά ένα ερωτηματικό έχει μπει, προφανώ αυτό ταλανίζει του Ευρωπαίου. Τρίτο γεγονό, πιο εσωτερικό αν θέλετε και συνδέεται πάλι με μια αντίληψη τη πραγματικότητα, είναι προφανώ το δημοψήφισμα για το Brexit, δεδομένου ότι επικράτησε η αντίληψη και αυτό ήταν πραγματι... πραγματικότητα εν μέρη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξερχόταν από, τις οργανώσεις, από την Οργάνωση για την Ασφάλεια και την Άμενα και πατούσε φρένο ως τώρα η Μεγάλη Βρετανία. Τώρα λοιπόν αυτό έχει σταματήσει και μπορούμε να συνεχίσουμε. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν σε δραστηριότητε, πρωτοβουλίε, σε μέσα και εργαλεία και προφανώ δεν πρόκειται να απαρνηθώ και να αρνηθώ την ε, σημασία του. Ε, όλα αυτά λοιπόν καλά και ωραία, αλλά δεν αρκούν σε καμία περίπτωση. Και αυτό που διαπιστώνω στην παρούσα φάση είναι το εξή. Αυτή η ορμή η οποία έχει σχηματιστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια σταδιακά μειώνεται. Γιατί διαπιστώνουμε ότι είμαστε αντιμέτωποι με κρίσει και όταν είμαστε αντιμέτωποι με κρίσει δεν είμαστε σε θέση να τι αντιμετωπίσουμε σωστά. Δεν έχουμε στο σωστό εξοπλισμό. Τα τρία αυτά στοιχεία όμω τα οποία ανέφερα, ιδιαίτερα τα δύο πρώτα, δεν πάβουν να υφίστανται και θα συνεχίσουν να μας ταλανίζουν. Να επισημάνω λοιπόν δύο στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και τρία στοιχεία τα οποία θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Καταρχάς, πιστεύω, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε σημαντικά έγγραφα, να καταρτίζουμε σημαντικά έγγραφα. Και πάλι μπορεί να σας κάνει λίγο εντύπωση που το λέω εγώ αυτό, αλλά πιστεύω κράτατα ότι δεν χρειαζόμαστε αυτό στην παρούσα φάση. Ασφαλώς, πάντα Καλό είναι να υπάρχουν κάποιες στρατηγικές πηξίδες, λευκές βίβλοι κτλ. κτλ. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά αυτά τα πράγματα παίρνουν πολύ χρόνο, πιστέψτε με. Και από πολλές απόψεις τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως το Συμβούλιο είναι πιο αρσενικά και όχι τόσο θηλυκά. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αν χρειαστεί να επιλέξουμε λοιπόν προτεραιότητες, να μην επικεντρωθούμε στην κατάρτιση περίπλοκων εγγράφων για να μπορέσουμε και να ταπανίσουμε τόσο πολύ χρόνο για να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες. Καλύτερα λοιπόν να επικεντρωθούμε σε άλλα θέματα. Και θα σας πω αργότερα σε τι πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεύτερο στοιχείο. Να μην ξοδέψουμε πολύ χρόνο, γιατί ήδη έχουμε χάσει χρόνο, για να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή συμφωνία για το ποιο είναι το νόημα και το έβρος της στρατηγικής αυτονομίας. Ε, για να σκεφτούμε δηλαδή αν σωστά κάνουμε και μιλάμε για αυτονομία, μήπως να μιλάμε για κυριαρχία, ευρωπαϊκή κυριαρχία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς, να συνεχίσουμε να το κάνουμε σε ό,τι αφορά την κατάρτιση της πολιτικής, όμως δεν πιστεύω ότι αυτό χρειαζόμαστε και αυτό πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Αυτά λοιπόν για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, δεδομένων και των συζητήσεων που λαμβάνω χώρα. Προσπαθούμε να βρούμε και έναν ορισμό μέσα σε όλα που θα αρέσει και στον ΟΗΕ. Στη ΕΠΑ, συγγνώμη. Γιατί αυτό έγινε το 2013. Τότε λοιπόν έγινε αποδεκτή. Αποδεκτό ορισμό αυτό. Πλέον είναι πιο αμφιλεγόμενο. Γιατί, γιατί δεν αρέσει στην κυβέρνηση Τραμπ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς, η κυβέρνηση Τραμπ δεν νοιάζεται δεν καθόλου για την ε, στρατηγική αυτονομία. Πολύ απλά δεν της αρέσει η ιδέα αυτή. Ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνάς ε, θα χρησιμοποιηθεί ο ΙΜΕ για την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Κλάδο Άμυνας. Αυτό δεν αρέσει στον Τραμπ. Δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο θα ορίσουμε την αυτονομία ή όχι. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τρία στοιχεία τώρα για το τι πρέπει να κάνουμε και εδώ θα κλείσω. Καταρχάς, συνοχή και συνεχτικότητα. όντω. υπάρχει αυτός ο μακρύς κατάλογος με όλα τα κρονήματα τα οποία εφαρμοστήκαν και πολλά από αυτά είναι λίγο ασάφη παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η εργασία και η δουλειά για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Υπάρχει ακόμα κάποια ασάφεια σε σχέση με το πόσο όλα αυτά δένουν και κλειδώνουν μεταξύ του σε στρατηγικό επίπεδο, κατά πόσον λειτουργούν ε, τα στοιχεία αυτά και με το βιομηχανικό σκέλος και το σκέλος των ικανοτήτων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λειτουργούν με συνεκτικό τρόπο. Είναι απαραίτητο και όλα αυτά να γίνουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, παράλληλα με την ανάπτυξη ικανοτήτων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και είναι σημαντικό να το πετύχουμε αυτό, γιατί πολλές από τις ικανότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν, όχι όλες, αλλά πολλές, σε βάση περιπτώσει, ουσιαστικά σκοπό έχουν να δρουν ως αποτρεπτικά και ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να δρά με τέτοιο αποτρεπτικό τρόπο και θα παραμείνει το να το απογνωρίζουμε. Υπάρχει λοιπόν το θέμα τη εσωτερική συνοχή μεταξύ των διαφόρων εργαλείων και των πολιτικών και των θεσμικών των θεσμών, αλλά και το εξωτερικό σκέλο, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεύτερο και πιο σημαντικό ενδεχομένω, το θέμα των χρημάτων. Αν μετά όλες τις μεγάλες διακηρύξεις και δηλώσεις Εξαγγέλουμε, προεξαγγέλουμε 30 δι ε, για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για την ε, άμυνα και τελικά καταλήξουμε μετά από όλε αυτέ τι ωραίε διακηρύξει να έχουμε τα μισά χρήματα στα πλαίσια του ΠΔΠ. Ειλικρινά θα γελιοποιηθούμε, πιστεύω. Το λέω έτσι ξεκάθαρα, δεν ξέρω πώ αλλιώ να το πω. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο όταν μιλάμε για την άμυνα, αν μιλάμε για στρατηγική αυτονομία, αν τα συζητάμε λοιπόν όλα αυτά, θα πρέπει να βοηθήσουμε το σκοπό μας. Και κατά τρίτον, και εδώ συμφωνώ α, απόλυτα με τον Πιέρ, στο λειτουργικό σκέλος και το έθεσες πραγματικά με απόλυτα σωστό τρόπο. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο επίπεδο της ανάλυσης της δράσης του έχει λάβει χώρα η δράση, όχι αντίστροφα. Και εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις όπου αυτό θα πρέπει πραγματικά να υλοποιηθεί. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να σκεφτούμε πιο πολύ το Ιράκ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ΙΠΑ στο Ιράκ είναι θέμα του πότε, όχι του αν θα αποσυρθούν. Το θέμα είναι πότε θα αποσυρθούν και πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ Θα ήταν φρικτή ιδέα να εμπλακεί στο Ιράκ για πολλούς λόγους. Πρώτος και καλύτερος είναι φυσικά η πολιτική κληρονομιά, η πολύ βαριά πολιτική κληρονομιά του ΝΑΤΟ στο Μέσα Ανατολή. Πολλά ωραία πράγματα έχει κάνει το ΝΑΤΟ, δεν λέω, και στην Ευρώπη κυρίω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη θέση στη Μέσα Ανατολή. Εκ παραλλήλου, οι Ιρακινοί χρειάζονται υποστήριξη. Και ζητούν υποστήριξη. Και του αρέσουν και οι Ευρωπαίοι. Έχουμε λοιπόν παρουσία με την πολιτική επιχείρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε αποστολές στρατιωτικής εκπαίδευσης. Φυσικά, τίθεται και το θέμα της ε, καταναγκαστικής ε, προστασία. Ακόμα και αν συμφωνήσουμε για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του Ιράκ, θα πρέπει να υπάρξει ε, υποχρεωτική προστασία. Αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, ανοιχτό εν πάση περιπτώσει, κλειστό θέμα είναι, για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και θα ήθελε να το κάνει αυτό. Εδώ λοιπόν ε, πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση κλειδί. Το ίδιο ισχύει και τη Λιβύη. Να φανταστούμε ενδεχομένω μια αποστολή εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με κάποια α, πολυεθνική αποστολή προστασίας. Αυτό θα ήταν μια περίπτωση πρακτική, όχι θεωρητική, όπου θα είχαμε μια ομάδα ευρωπαϊκή η οποία θα δρούσε παράλληλα με κάποια άλλη τέτοια δύναμη. Και φυσικά, ίσως πιο σημαντικό, πιο σημαντικό για το Ιράκ παρότι υπάρχουν θέματα, υπάρχει ο κίνδυνος εκεί της, ανά, της επανεμφάνισης του ISIS. Πιο σημαντικό θέμα λοιπόν είναι η Λιβύη. Η ΙΠΑ μπορεί να, το, να μας αρέσει, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εμπλακούν στην Λιβύη, το είπαν, το ξαναείπαν, μας έκαναν να το καταλάβουμε. Η όλη πορεία της κατάστασης δείχνει ακριβώς την απουσία των ΙΠΑ στην Λιβύη. Αυτό είναι. Αν δεν εμπλακούν οι ΙΠΑ, αν δεν εμπλακεί η Ευρώπη, αυτοί που θα εμπλακούν, που είναι φανερό, δεν νομίζω ότι θα εμπλακούν προς όφελός μας. Το θέμα λοιπόν είναι και πάλι ένα θέμα που βασίζεται στο εξή. Θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο ή όχι. Και αν θέλουμε, η Λιβύη είναι η καλύτερη περίπτωση. Και άλλη περίπτωση όπου είναι δύσκολη, περίπλοκο, χωρίς ασφάλειες, περιβάλλον, απαιτεί ευρωπαϊκή παρέμβαση, αλλά αν δεν δούμε κάτι τέτοιο την επόμενη πενταετία, θα είναι περιττό, για να μην πω βλαβερό, να έχουμε νέα κείμενα. Ευχαριστώ. Μπρουκστίγνερ. Προσπαθήστε κι εσείς, το λέω και το ξαναλέω, να μην μιλήσετε πάνω από 10 λεπτά. Πρέπει να έχουμε ένα διάλογο, όχι πέντε απλά διαλέξεις. Και γι' αυτό θα έχουμε μια τελευταία παρέμβαση και στη συνέχεια ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Στίγνερ. Um, Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, είναι ασυνήθιστο να είμαι εδώ πάνω στο Προεδρείο. Συνήθω είμαι στο βάθο τη έκθεση και καλύπτω αυτά που λένε οι υπόλοιποι. Ε, από τη στιγμή που παρακολουθώ την επικαιρότητα. Θα κάνω ό,τι μπορώ όμω. Νομίζω ότι πρέπει να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Ε, κάποια ε, που σκέφτηκα όταν διάβασα αυτό το ενημερωτικό σημείωμα και να απαντήσω ε, και σε ορισμένα ερωτήματα των ομιλητών. 30 χρόνια καλύπτω το ζήτημα. Είμαι απεσιόδοξο. Θα μου άρεσε να ήμουν αισιόδοξο, αλλά είμαι απεσιόδοξο ω προ του φιλόδοξου στόχου τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα η ε, ολοκληρωμένη ενιαία προσέγγιση, ε, ε, ενιαία πολιτική, ωραία λόγια αυτά. Αρέσουν στην Ευρώπη τα ωραία λόγια, αλλά σε πολύ λίγα μέρη μια πραγματικά ολοκληρωμένη και ενιαία προσέγγιση έχει κομίσει αποτελέσματα, ίσως με την εξαίρεση των Βαλκανίων που είναι η πίσω αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μπλακεί ποτέ σε σκληρούς στρατιωτικούς στόχους, δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, και να έχει οικονομική ανάπτυξη και πολιτισμική ας ανάπτυξη σε μια ζώνη εμπόλεμη. Στο Μαλί, στην Πουρκίνα Φάσο. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Να είμαστε πιο μετροεπαθείς για το ρεαλισμό των προσδοκιών μας και να παραδεχόμαστε κατά πόσο είναι εφικτή αυτή η προσέγγιση και να μην κρεμάμε αυτό το καρτελάκι, αυτή την ταμπελίτσα σε οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ακούγεται ωραία. Να το πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή είναι μια αποστολή αντιτρομοκρατική από εκεί και τίποτα άλλο και δεν αποτελεί μια, ε, μέρος μιας ε, πιο ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης, γιατί αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Άρα μένουμε στην αντιτρομοκρατική δράση, π.χ. και σε τίποτα άλλο. Αυτό καταρχάς. Ε, το έγγραφο για το θεσμικό ε, πλαίσιο προτείνει το QNV. Πράγματι πρέπει οι βουλευτές να ασκήσουν πίεση στο Συμβούλιο να ε, κινηθεί προς το QNV. Το θέμα είναι ποιος, έκανε, ποιος ήταν πρώτος, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό τη κότα. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους θέσεις, αλλά όταν δεν πρέπει να συγκλίνουν, αλλά αν συγκλίνουν τελικά θα συμβεί μία φορά στη ζωή μας και τότε δεν θα έχουμε QNV να βασιστούμε, ενώ θα έχουμε σύγκληση. Πρέπει να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, πού να το εφαρμόσουμε σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν ξέρω αν είναι αυτή η σωστή άγουσα, αλλά... Ακόμα και αν αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας πάρει το QNV και συνεδριάσει πριν το πραγματικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής, ε, πάλι ε, δεν θα είναι αποτελεσματικό. Τώρα για το έγγραφο για το TDIB, Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μέγερ, 100% όσα ε, χρήματα να έχει κανείς και για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και για τις λοιπές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ήδη υφιστάμενες ή τις μελλοντικέ δεν θα αλλάξει το TDIP, ακριβώς διότι κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει να χάσει. Μας αρέσει η έκφραση win-win, αμοιβαία υποφελή κατάσταση, αλλά είναι ελάχιστες οι καταστάσεις που είναι αμοιβαία υποφελής. Κανένα κράτος μέλος δεν θέλει να χάσει, να αποδυναμώσει το δικό του αμυντικό σκέλος για το ευρύτερο ευρωπαϊκό καλό. Ε, έξι διαφορετικά σώματα επιτρόπων έχω παρακολουθήσει να το λέμε, είναι έξι διαφορετικές θητείες επιτρόπων, αλλά, αλλά δεν αλλάζει, όλοι το γνωρίζουν. Και τώρα δύο λόγια για τη στρατηγική αυτονομία και παραμένω σύντομο γιατί πράγματι είναι δίκαιο εσεί οι βουλευτέ να υποβάλλετε ερωτήσει και να μην μονοπολούμε εμεί το μικρόφωνο. Στρατηγική αυτονομία τι σημαίνει ότι ε, ε, τελικά να υπερασπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον εαυτό τη στρατηγικά και στρατιωτικά, να καταφέρει εκεί να φτάσει, κάτι το οποίο δεν μπορεί να πράξει. Α το θέσουμε κατά μέρο. Α μιλήσουμε για μια πιο καλοήθη εκδοχή του, ε, για την ε, καλοήθη ε, εκδοχή της στρατηγικής αυτονομίας, ε, για παράδειγμα, στον εφοδιασμό, στην επιμελητία ή σε συγκεκριμένες δράσεις. Και ούτε αυτό έχετε. Αφού δεν το έχετε, ε, να μιλήσουμε για αποφάσεις, ε, για να είναι ισχυρές οι αποφάσεις πρέπει να υπάρχει ισχυρό γεθά εδώ στις Βρυξέλλες, ευρωπαϊκός αν θέλετε, ε, γενικό επιτελείο που να μπορεί να είναι πραγματικά ενιαίο και να μπορεί να λάβει ισχυρές αποφάσεις γρήγορα και να υπάρχει δημόσια βούληση από τους πολιτικούς μας ηγέτες να αφήσουν ε, ε, Ευρωπαίους στρατιώτες να πεθάνουν επιτόπου στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι ταμπού όμως. Δεν μπορεί όμως να έχει κανείς στρατηγική αυτονομία χωρίς να έχει αυτή τη βούληση και μάλιστα δημόσια προκειμένου να πετύχει το στόχο. Άρα είναι παραπλο... παραπλανητικό προς τους πολίτες και εγώ είμαι Βέλγος πολίτες να δίνουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζει στρατηγική αυτονομία ενώ δεν το πράττει τελικά. Και ε, Ίσως χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση, μια νέα έκφραση για αυτή την έννοια, γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν το εφαρμόζουν. Δεν πρόκειται να έχουμε στρατηγική αυτονομία παρόλο που τη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα και παρόλο που ξέρω ότι δεν σα αρέσουν οι νέε λέξει, ίσω πρέπει να εφεύρουμε ένα νέο όρο και όχι στρατηγική αυτονομία για να μην παραπλανούμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Ξέρω ότι τάραξα τα νερά, αλλά θα ολοκληρώσω κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Η κυρία Νόημαν έχει το λόγο. Ο κύριο Μέγερ εκτό μικροφώνου. Ο κύριο Γκάλερ εκτό μικροφώνου. Ναι, θα σα δώσουμε το λόγο, λέει η πρόεδρο. Όλοι, πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο, θα τον πάρετε όλοι το λόγο. Ε, η κυρία Νόημαν, καταρχά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Τίκνερ, αλλά και του υπολείπους. Ε, ήταν οι ομιλίες σας πολύ ζωντανές, πολύ παραστατικές, πολύ έντονες. Ε, ήταν και αφιλεγόμενες με την έννοια ότι υιοθέτησαν διαφορετικές απόψεις. Ε, Καλό είναι αυτό. Δύο είναι τα ζητήματα που θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, η σχέση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς αυτά. Βλέπουμε διαφορετικές έννοιες να επικρατούν σε διαφορετικές χώρες. Πριν από δύο χρόνια, ε, για το θέμα της Λιβύης, ε, τα κράτη-μέλη κινούνταν προς διαφορετικές και μετά έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα έννοια της ε, κοινή ε, πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και τελικά δίνεται εντολή σε ένα κράτος μέλος να προχωρήσει αυτό που ε, είναι η μέθοδος Μπαρνιέ με το Brexit, όπου αυτός ε, μίλησε εξ ονόματος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα μπορούσε και αυτή να είναι επιλογή για τις αποστολές της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, να προχωρήσουν οι λίγες χώρες, ενώ άλλες δεν θέλουν να προχωρήσουν. Εξίσου βλαβερό είναι να έχουμε μια μικρή ευρωπαϊκή αποστολή και μετά να έχουμε πολύ μεγάλες συνεισφορές των κρατών μελών παράλληλες στη συμμαχία αυτών που θέλουν ή στην ε, Βορειοατλαντική Συμμαχία και τελικά το είδαμε αυτό και στο Μαλί να παρακολύουν ε, αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Μέση Ανατολή Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών στη Σαουδική Αραβία χθε και μου είπε ότι εμεί προτιμούμε τι διμερείς συνομιλίε. και με αυτό το χάσμα και αυτό το χάο, εκεί θα επιστρέψουμε στη διμερή προσέγγιση και για τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό. Είπατε να εκεί αυτά τα οποία επιθυμούμε, ε, αυτά να χρηματοδοτούμε. Αλλά όταν επιθυμούμε και εκφράζουμε αυτές τις επιθυμίες, να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας. Ε, θα πρέπει ε, να κάνουμε πράγματα μαζί και όχι να ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσει περισσότερα γιατί τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να παραχωρήσουν ε, κυριαρχία. Γιατί αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά, είναι ε, σοβαρά πράγματα της κακιάς ώρας. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ε, από εκεί και πέρα. Πιστεύετε ότι ε, δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξία γιατί δεν υπάρχει βούληση ή γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη επάρκεια, εξοπλισμό, δεν, υπάρχουν, δεν δυνάμεθα ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ο κύριος Γκάλερ, γιατί δεν θέλει κάποιος άλλος γιατι δεν θελει καποιος αλλο συντονιστη στο λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω να πω προς την κυρία Τότσι. το εξή. Συμφωνώ ε, με αυτό που είπατε. η σημερινή ε, κυβέρνηση είναι αυτή η οποία δεν καταλαβαίνει ε, πού στοχεύουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές αμυντικές προσπάθειες. Η προηγούμενη το είχε καταλάβει. Ναι, χρησιμοποιούμε τα δικά μας χρήματα για τη δική μας βιομηχανία και αυτό είναι εξωφρενικό βεβαίως. βεβαίως. Ωστόσο, λέτε ότι δεν θα πρέπει να παραχθεί άλλο ένα μεγάλο έγγραφο μακροσκελές. Προσθέτω κόμμα που δεν περνάει από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και άρα δεν ρωτήθηκαν τα κράτη-μέλη για τη συνδιαμόρφωσή του και γι' αυτό δεν θεωρούν την Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική ως δικιά τους Ευρωπαϊκή Παγκόσμια Στρατηγική. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος που συνέβη τότε. Δεν πέρασε το κείμενο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για να το προσυπογράψουν, να το διαμορφώσουν. Τους σερβιρίστηκε και τα κράτη-μέλη δεν το κατάπιαν ως δικό τους προφανώς. Πρέπει να προσδιορίσουμε το δικό μας σε επίπεδο φιλοδοξιών. Πρέπει να μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες και για να φέρουμε σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την πορεία τα κράτη-μέλη, χρειαζόμαστε λευκή βίβλο για την ασφάλεια, έτσι ώστε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν σε αυτούς τους στόχους και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας στη συνέχεια, τις ε, στρατιωτικές και αμυντικές. Αναρωτιέμαι, συμφωνείτε με την άποψή μου την εξής, Πολλέ από τι πολιτικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί και σα θυμίζω και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013. Τα πρώτα δύο σημεία της ημερήσια διάταξης ήταν, ε, ε, είχαν να κάνουν με αμυντικά θέματα. Έτσι έγραφε η ημερήσια διάταξη. Υπάρχει ασφάλεια στην, ε, στον εφοδιασμό. Αυτό θαύτηκε κάπου. Γιατί. Και εμεί έπρεπε να πιέσουμε για το πιλωτικό πρόγραμμα και να υπάρξει μια πρώτη γραμμή του προπολογισμού για τέτοια θέματα. Και τελικά κάπου οδήγησε αυτή η προσπάθεια για την οποία και είμαστε περήφανοι. Επίσης, η στρατηγική αυτονομία πρέπει να τύχει ορισμού, πρέπει να την ορίσουμε. Υπάρχει στην νομοθεσία για το αμυντικό ταμείο, άρα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει στρατηγική αυτονομία με τρόπο κατά τον οποίο να λέει ότι ε, πρέπει να είμαστε σε θέση να δράσουμε εάν π.χ. η προσφυγή σε πόρους του ΝΑΤΟ δεν είναι εφικτή. Μπορεί να υπάρχει κάποιο βέτο. Να θέλω εγώ να κάνω κάτι στη Λιβύη και να μην εξαρτώμαι από τους Ρώσους ή τους Τούρκους. Γιατί δεν νομίζω ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντά μας. Ενώ π.χ. μπορεί να είναι η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ. Ε, δεν εκπροσωπούν τα συμφέροντά μας και μπορεί να θέλουν δεν, πρέπει να πρέπει εμείς να καθόμαστε να περιμένουμε να προλαβαίνουν τις εξελίξεις οι Ρώσοι ή οι Τούρκοι. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Αυτή είναι η επιστολή του κυρίου Μπορέλ. Ε, θα πάρουμε απάντηση. Νομίζω ότι παίρνουμε απάντηση μέσα σε 100 μέρες από κάθε επίτροπο. Τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Νομίζω ότι αν οριστεί θα προχωρήσουν τα πράγματα και θα καταλήξουμε σε καλό ορισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπασέσκου παρακαλώ. I heard today one... Δόξα τω Θεώ, κατάλαβα τι θα πει στρατηγική αυτονομία. Δεν είναι ότι δεν σημαίνει τίποτα. Δεν έχουμε περιεχόμενο για την έκφραση αυτή. Και δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αυτόνομοι αυτή τη στιγμή και για μεγάλο διάστημα κατά πάσα πιθανότητα. Η στρατηγική αυτή αυτονομία είναι δημιουργία like, όπως αυτές τις κυρίας που μας κρατάει σε μεγάλες ομιλίες. Δεν είμαστε αυτόνομοι γιατί δεν έχουμε πυρηνικό οπλοστάσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η ανάλυση μου μάλλον από την εμπειρία που έχω ως πρόεδρος. Δείτε τους Ρώσους. Έχουν μία η οικονομία μικρότερη από της Ιταλίας, αλλά είναι υπερδύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε κομμάτι της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης ή όχι. Αν θέλουμε να είμαστε μέρος αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις. Αν ναι, θα πρέπει με τον α ή β τρόπο να μείνουμε εταίροι τον ΙΠΑ προς το παρόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Οι παίκτες στην Ευρώπη σήμερα είναι η Τουρκία και η Ρωσία. Κανείς μας ρώτησε. Προσπαθήσαμε να το παίξουμε διαμέσου στην Ιρανοαμερικανική διένεξη. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την διαμεσολάβησή μας. Ας είμαστε ειλικρινεί, Όταν μιλάμε για τις δυνατότητές μας να γίνουμε μεγάλοι παίκτες, Έχω την άποψη ότι με τον α ή β τρόπο πρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μείνουμε εταίροι με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Έστω και αν οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν τον Τραμπ ως ε, πρόεδρο. Δείτε την αριστερή πτέρυγα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όταν ε, έγινε η εισβολή στην Κρυμαία, όλες οι πρώην κομμουνιστικές χώρες ε, ανησύχησαν. Ξέχουμε την εμπειρία. Οι Ρώσοι απλώς περνάνε τα σύνορα. Και μπορούν να περάσουν τα σύνορα της, των κρατών της Βαλτικής ή της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας όπως έκαναν με την Ουκρανία. Αυτό δεν θα συμβεί διότι προς, προς το παρόν, διότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αποφάσισε να εγκαταστήσει αμερικανικό εξοπλισμό που είναι πλέον ε, εξοπλισμός του ΝΑΤΟ. Δεν είναι στη Ρουμανία, δεν είναι Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί στρατιωτικοί. Οι Αμερικανοί ήρθαν. Έφεραν 2.000 στρατιώτες με στρατό, με αεροπλάνα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εξαρτιόμαστε από τους Αμερικανούς για την ασφάλειά μας. Το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πυρηνικό οπλοστάσιο για να εξισορροπήσουμε την κατάσταση με, την, με τις Ηνωμένες τη Ρωσία, την Κίνα, το Πακιστάν, την Ινδία είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Ευρώπη σήμερα. Άρα η μόνη λύση που υπάρχει είναι να συνεχίσουμε να είμαστε εταίροι των Ηνωμένων και μαζί να προσπαθούμε να μπούμε στο παγκόσμιο παιχνίδι. Γιατί δεν έχουμε στρατιωτικές ικανότητες. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να κάνουμε τις αποστολές μας στην Αφρική. Εκεί έχουμε τεράστια ιστορική ευθύνη για την Αφρική. Κάποιοι από εμά τουλάχιστον. Είναι γείτονέ μας στη μεσο, από την νότια πλευρά της Μεσογείου. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην Αφρική. Δεν έχουμε όμως το θάρρος να το κάνουμε αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ. Chris Πέτερς. Να πω στον κύριο Μπασέσκου ότι κάποιες, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν και θάρρος να είναι στην Αφρική και χάνουν και ζωές εκεί. Όχι αρκετές δυνάμεις για μη είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο εγκρίναμε μία έκθεση για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής της ε, αμυντικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας όπου δίνουμε έναν σαφή ορισμό για την ανάγκη να αναπτύξουμε μία ευρωπαϊκή στα, στρατηγική αυτονομία. Επίσης το διαβάσετε, Το ενέκριναν όλες οι ομάδες. Να είμαστε σαφείς. Το διαβάσετε κι εσείς ελπίζω. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Όταν συζητούμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία, να διαβάζετε τι έχουμε εγκρίνει. Κάποιοι δεν το ενέκριναν. Καλά. Αλλά υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία. Δεύτερον, ο κόσμος αλλάζει γρήγορα και συμφωνώ ότι η Ευρώπη τώρα πρέπει να αρχίσει να παρουσιάζει αποτελέσματα. Τι μπορεί να κάνει, τι θέσεις έχει σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο καινούργιο. Και το είπαμε. η γεωπολιτική αντίληψη των ΗΠΑ αλλάζει και άλλα πράγματα αλλάζουν. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν ήμουν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο Βέλγιο, το είχαμε πει. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, όχι ταπεινόφρονες. Εμείς είμαστε ταπεινόφρονες γενικά στο Βέλγιο γιατί είμαστε μια μικρή χώρα αλλά πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα για τον κόσμο. Δεύτερον, δεν θέλουμε μήνες και χρόνια συζητήσεων. Αλλάζει ο κόσμος. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε και εμείς μεταξύ μας ποια είναι η δική μας άποψη. Τι όραμα έχουμε για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον που είναι νέο. Αυτό είναι το βασικό για μας. Τι θέλουμε. Καλά. Εντάξει τις αξίες. Αλλά στη Real πολιτική, τι θέσεις έχουμε. Όταν έρχονται και λένε κάντε κάτι Ευρώπη ο κόσμος. Τι μπορούμε να κάνουμε. Χρειαζόμαστε αποστολές και στρατιωτική δράση. Και όταν δεν είναι δυνατό σε πέντε χρόνια να μην έχουμε πρόοδο. Δεν μπορεί σε πέντε χρόνια, αν δεν πετύχουμε κάτι τέτοιο, να έρθει ο νέο πρόεδρο Επιτροπή και να πει θα είμαστε γεωπολιτική επιτροπή. Αν δεν έχουμε κάνει κάτι την επόμενη πενταετία, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει. Δεν μπορούσαμε να πείσουμε άλλους, άλλες χώρες, άλλο κόσμο, ότι η Ευρώπη κάτι υποστηρίζει τέλο πάντων. Πριν δώσω το λόγο στους τέσσερις προσκεκλημένους μας, για να απαντήσουν. Να μιλήσω κι εγώ λίγο. Πρόεδρος είμαι στο κάτω-κάτω. Για κάποια από αυτά που άκουσα, τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε ή όχι μια στρατηγική πηξίδα. Δημιουργήσαμε έναν λαμπρό μηχανισμό αλλά είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε αν δεν εξηγούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Σήμερα η Κίνα έχει μια στρατηγική. Την ξέρουν όλοι. Την όρισαν, την εξήγησαν, την ξέρουν. One Belt, One Road κτλ. Και όλοι μπορεί να πούν, συμφωνούν, διαφωνούν, είμαστε υπέρ, είμαστε κατά. Η Αμερική έχει ένα σλόγγαν τουλάχιστον. America First. Και αυτό το καταλάβαμε. Όλα ακόμα και για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, από εκεί περνάνε. Εμείς έχουμε κάτι ακρονίμια. Δεν δημιουργήσαμε πολιτική βούληση στον τομέα της άμυνας. Ωστόσο, το είδαμε και στην, στην προεκλογική εκστρατεία, ότι όλοι οι πολίτες παντού λένε «Ευρωπαϊκή άμυνα». Αν δεν το δούμε ουσιαστικά, όχι μόνο δεν υλοποιούμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά καταβαραθρώνουμε ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως, τρέχουν από πίσω μας οι κρίσεις, ο κόσμος. Κάτι σαν το ζουρδέν κάνουμε. Κάνουμε πολιτική χωρίς να το ξέρουμε. Αλλά αν δεν το πούμε εμείς οι αιρετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων, ποιος θα το πει. Δεν είναι ότι ζούμε σε μια φούσκα. Υπάρχει, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που ζητούν άμυνα στην Ευρώπη. Πολλά είπα. Ξαναδίνω το λόγο στους ομιλητές μας από το τέλος προς την αρχή. Επτά λεπτά ο καθένας. Έφυγε η κυρία που έθεσε το θέμα αυτό. Για το κατά πόσο να μπορούμε ή δεν θέλουμε να δράσουμε σε ό,τι αφορά τους ε, κρατικούς φορείς και το συζητούσαμε και με τον επικεφαλής ε, του IEA και συμφώνησε σε ό,τι αφορά τα θέματα τη αυτονομία, Είπε ότι πρέπει καταρχά να κοιτάξουμε το θέμα τη ικανότητα, γιατί το θέμα τη προθυμία και τη βούληση δεν υπάρχει ακόμα και υπάρχει μια εγγενή ε, απροθυμία σε όλε τι πρωτεύουσε να μεταφέρουν πιο πολλέ αρμοδιότητες στι Βρυξέλλε. Είναι γεγονό αυτό, αλλά θα πρέπει να το αποτεχτούμε. Τα επόμενα 5-6 χρόνια Ενδεχομένω θα πρέπει να αφιερώσουμε όλε τι προσπάθειέ μα για να αναπτύξουμε τέτοιε ικανότητε. Γιατί οι Ιταλός, οι Ευρωπαίοι, οι ηγέτε διαρκώ λένε «Α, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά γιατί δεν υπάρχουν ικανότητε. Ε, θα του πούμε «Υπάρχουν πλέον ικανοτήτε και θα πρέπει αυτή να γίνει η ε, μεταφορά των αρμοδιοτήτων». Η κυρία Τότσι, να απαντήσω εν συντομία για το θέμα των πρώτων μελών. Ακούσαμε και το παράδειγμα της Λιβύης. Προφανώς, ναι. Γι' αυτό υπήρχε ως τώρα α, αδράνεια. Αυτό που είναι ενδιαφέρον ωστόσο είναι το εξή, ότι αυτό που ενδεχομένως να αλλάξει τώρα, υποαίρεση δεν είμαστε βέβαιοι, αλλά μπορεί και να αλλάξει από ένα κράτος μέλος υπήρξε μια μετακίνηση. Είναι τελικά και πιέρνει από το άλλο άκρο. Αυτό που αλλάζει όμως είναι το εξής. Συμφωνούν ότι οι διαφωνίες τους είναι πιο περιορισμένες από ότι η συμφωνία τους ότι δεν θέλουν η Ρωσία και η Τουρκία να βρεθούν τελικά να κανονίζουν και να κινούν τα νήματα. Θα πρέπει να επαναξιολογηθεί λοιπόν η σχετικότητα των όποιων διαφορών έχουμε στις αντιλήψεις μας. Και συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι αφορά το θέμα του να δοθεί εντολή στα κράτη-μέλη. Ιδανικά δεν θα έπρεπε να έχει την εντολή αυτή μόνο ένα κράτος μέλος, θα έπρεπε να είναι μια ομάδα κρατών μελών, γιατί θεωρώ ότι αυτό τελικά καθιστά τις ομάδες επαφής ένα υγιή μια ομάδα εργασίας που θα έχει θεσμική σύνδεση με το σύνολο των θεσμών, όπου θα υπάρχει ευελιξία, ταχύτητα αντίδρασης, χωρίς όμως τα μειονεκτήματα τα οποία είναι η έλλειψη νομιμότητας και φυσικά και η διέρεση αν ε, όλα αυτά συμβούν τελείως ανεξάρτητα από το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων ε, συμφωνώ. Εκ παραλίλου, όμως θέλω να τονίσω το θέμα αυτό της απροθυμίας, γιατί όντως δεν έχουμε την ικανότητα σήμερα να ξεκινήσουμε μια μεγάλη απόστολη και επιχειρήση. Δεν έχουμε τη στρατηγική αυτή ικανότητα. Όλα αυτά τα οποία τα θέλαμε το 2013 εξακολουθούμε να μην τα έχουμε. Αυτό στέκει. Αλλά για να κάνουμε αυτά που συζητάμε εδώ και τώρα, στο Ιράκ στη Λιβύη. Έχουμε, έχουμε πραγματικά τις ικανότητες να τα κάνουμε αυτά. Άρα, είναι θέμα προθυμίας και θα πρέπει να αποδεχτούμε και τους κινδύνους ότι ενδεχομένως να υπάρξουν θύματα. Αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο. Αυτή λοιπόν η προθυμία θα εξακολουθήσει να υφίσταται όσο ε, ζούμε στην ψευδέστηση ότι κάποιος άλλο θα έρθει, κάποιος άλλος δηλαδή είπα, έχουν όνομα, θα μας ε, φροντίσουν. Είμαστε σε μια πλάνη, σε ένα όνειρο απατηλό και θεωρούμε ότι ο Τραμπ είναι το πρόβλημα. Και πολύ φοβάμαι, κυρίε και κύριοι, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Τραμπ. Υπάρχει πιο δραστατικό πρόβλημα και θα λάβει διαφορετική μορφή στο μέλλον, αλλά ουσιαστικά οι ΙΠΑ ΕΕ έχουν μία στρατηγική πρόκληση, μία και μεγάλη, και αυτή δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε η Μέση Ανατολή. Το όνομά τη είναι Κίνα. Και προφανώ όλοι έχουν περιορισμένου πόρου και άρα μοιραία. Εκεί θα εστιάσει τις προσπάθειές της, σε αυτή την προτεραιότητα. Αυτή λοιπόν η προθυμία θα ξεκινήσει τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Τώρα είμαστε ακόμα στην ψευδέστηση ότι έχουμε εναλλακτικέ λύσει. Και μην με παρανοήσετε, δεν είμαι κατά των λευκών βίπλων, των εγγράφων κτλ. Αυτό που λέω είναι το εξή. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο και περιορισμένου πόρου Καλά θα κάναμε να δαπανίσουμε το χρόνο που έχουμε για να πετύχουμε μία συμφωνία. Από να πετύχουμε μία συμφωνία, να πετύχουμε και να καταφέρουμε να κάνουμε κάτω. Είδαμε και τι έγινε το 2013 με την ε, η διεκτησία των εγγράφων από πλευρά του Συμβουλίου και πόσο καιρό πήρε. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Άρα, α μην ταπανίσουμε πάρα πολύ χρόνο στη θεωρία, ιδιαίτερω γιατί αυτό το χρόνο το χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτά που πραγματικά πρέπει να γίνουν. Να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιμό. Ευχαριστώ και εν συντομία γιατί λίγο πολύ τα είπαμε αυτά που χρειάζεται να πούμε. Δύο-τρία σημεία να προσθέσω και εδώ θα διαφωνούσα θα έλεγα με κάποιους από τους ομιλητές μας. Καταρχάς, πρώτο σημείο, σε όλο τι αφορά το όλο θέμα του κατά πόσον είμαστε πρόθυμοι ή κατά πόσον δεν έχουμε τις ικανότητες και τα δύο. Αλλά από την άλλη να σας πω δεν είμαι και τόσο απεσιόδοξο. Αντίθετα, με τον κύριο αυτό που βλέπουμε είναι το εξής αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ όλων των κρατών μελών, κάποιοι που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις μπορούν να συνεχίσουν μόνοι τους. Αυτό το ονομάζουμε ευελιξία. Το έχουμε συμφωνήσει και αυτό συμβαίνει και στην πράξη. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό θεωρώ προσωπικά είναι το εξή. Μέσα σε αυτό το νέο ευέλικτο μορφότυπο που επινοούμε, τουλάχιστον να φροντίσουμε με τακτικό τρόπο να περιληφθούν ή τα θεσμικά όργανα. Γιατί ένα από τα επιτεύγματα που καταφέραμε να πετύχουμε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν το GCPOA. Και αυτό το πέτυχαν τρία κρατημέλη, μόνο τους. Με την υποστήριξη όλων των υπόλοιπων βέβαια, γιατί είχαμε την ύπατη εκπρόσωπο η οποία ε, συμμετείχε. Αυτή την πρακτική λοιπόν την έχουμε χάσει και κακώς ε, τη χάσαμε να επανέλθουμε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα στην Ουκρανία με την διαδικασία του Μίντς και εγώ το έλεγα πάντα ότι ε, με λυπούσε το γεγονός ότι δεν συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιμο ακόμα και τώρα. Αλλά τέτοιου είδους νοοτροπία ε, χρειαζόμαστε για να ξεπεράσουμε αυτή την απεσιοδοξία που ε, μας μαστίζει στην παρούσα φάση. Υπάρχει λιγμού για όσους θέλουν να προχωρήσουν προς τα εμπρό. Και γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, να πω και δύο λόγια για το QMV. Εγώ υποστηρίζω όπως και όλοι μας, την ε, ειδική πλειοψηφία. Δεν είμαι βεβαίως ότι για την πολιτική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας αυτό βγάζει νόημα. Σκεφτείτε το. Και αυτό για το τμήμα τη πρόταση που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκεφτείτε λοιπόν, όταν συζητάμε θέμα κυρώσεων, αν αποφασίσουμε να επιβάλλουμε ειδική πλειοψηφία. Όσοι έχουν καταψηφίσει, τι θα κάνουν. Φυσικά θα του πούμε ότι είναι να σεβαστείτε την απόφαση τη πλειοψηφία. Αλλά θα πούνε, θα συμφωνώ και πολύ απλά θα πάω και θα κινηθώ μόνο μου. Έχουμε τέτοιε περιπτώσει, όπω είδαμε με το όλο ε, σχέδιο ε, με την εγκατάσταση στην ομάδα Visegrad που ασκεί πιέσει και θα βρεθούμε σε τέτοιε θέσει στην πολιτική εξωτερικής, εξωτερικών υποθέσεων, στην πολιτική ασφάλεια. Φαντάζεστε τι μα, καταστροφή θα σήμαινε αυτό, τι είδου μήνυμα θα απέστελε, απέστειλε. Εδώ λοιπόν θα συστήνα προσοχή, να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Τελευταίο θέμα, είπα και να το. Κύριε Πρόεδρε, σε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, πραγματικά διαφωνώ μαζί σας σε ό,τι αφορά την πυρηνική ε, το απερινικό αντικίνητρο. Εκεί φαίνονταν τα πράγματα πολύ επικίνδυνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελέσει ενδιάμεσο. Πιστεύω ότι υπάρχουν όλοι οι τρόποι να αντιμετωπίσουμε την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αποσυρθεί από την πυρηνική συμφωνία. Το έχουμε κάνει και το έχουμε κάνει με διαφορετικού τρόπου στο παρελθόν. Το 82, όταν η κυβέρνηση την ΕΠΑ ήθελαν οι Ευρωπαίοι να μποϊκοτάρουν τον αγωγό αερίου με τη Σοβιετική Ένωση και καταφέραμε να προχωρήσουμε. Το ξεκαθαρίσαμε παρά την αντίσταση τον είπα. Φυσικά έχουν αλλάξει και δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιε συγκρίσει, εδώ συμφωνώ, αλλά ενδεχομένω να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να καταδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό διαμεσολαβητή. Έχουμε, έχουμε και καμιά φορά μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε στα οικονομικά ζητήματα. Να το σκεφτούμε όμω Τελευταίο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω. Όταν συζητάμε για τη ΣΥΠΑ και την αλλαγή στην πολιτική. Η στρατηγική αυτονομία ότι δεν είναι ε, δυνατή και θα πρέπει να μείνουμε στο ΝΕΤΟ. Ένα από τα πρόβλημα που με συναρπάζει είναι το εξή. Αυτό που βλέπουμε στην παρούσα σε, για παράδειγμα στο Σαχέλ, όπου προσπαθούμε να καταρτήσουμε ενός είδους στρατηγικής αυτονομίας. Και αυτό που βλέπουμε είναι ένας από τους βασικούς μας συμμάχους, οι Αμερικάνοι μας λένε ότι θα σας αφήσουμε σε ξύλους, μόνο σας. Μα το ΝΑΤΟ τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετεί αν δεν μπορέσουμε αν δεν μπορούμε να, συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε ότι είμαστε σύμμαχοι και ότι θα πρέπει να άλλο υποστηριζόμαστε. Και γιατί το και από την άλλη. Λέμε πάντα ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μείνουν στο ΝΑΤΟ. Αλλά κάποιοι από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει και αυτοί να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Η Νάταλη ανέφερε την περίπτωση του Ιράκ, όπου το θέμα της αμερικανικής απόσυσης δεν είναι θέμα ε, του αν, είναι θέμα του πότε. Και αυτό πραγματικά προκαλεί έκπληξη σε ό,τι αφορά την διατλαντική αυτή συμμαχία. Έτσι την θεωρούμε. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε λίγο πιο πολύ την στρατηγική αυτονομία, γιατί σε τέτοιου είδου καταστάσει ενδεχομένω να βρισκόμαστε όλο και πιο πολύ στο μέλλον. Και σε τελική ανάλυση, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται, είμαστε μόνοι μα σε θέση να τα προασπίσουμε. Αν μα εγκαταλείψουν οι σύμμαχοί μα, είμαστε σε θέση να προασπιστούμε τα συμφέροντα αυτά. Αυτό είναι το θέμα θα πρέπει να δοθούν να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά. Ίσως όμως εμείς τελικά θα αφήσουμε τους συμμάχους μας, κυρία Πρέσβη, στο Αφγανιστάν στο Ιράκ. Ο κύριος Μάγερ, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια για το θέμα του κατά πόσο δεν είμαστε καλά εξοπλισμένοι ή δεν έχουμε βούληση. Εξαρτάται από την αποστολή. Υπήρξαν αποστολές που δεν υπήρχε πολιτική βούληση, αλλά είχαμε καλό εξοπλισμό. Και υπήρχαν περιπτώσεις όπου τα στρατεύματα ε, ε, υπήρχαν επί, επί χάρτου μόνο. Δεν θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε και να τα αποφασίζουμε. Εξαρτάται δηλαδή από την περίπτωση. Και επιστρέφω σε αυτό που είπε ο Πιέρ για την οτροπία το ότι μαθαίνουμε κάνοντας πράγματα, οργανώνοντας αποστολές, ότι με την πράξη έρχεται η πείρα. Συμφωνώ με αυτή την άποψη γενικά. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η συζήτηση είναι το εξής. Το κόστος της μη δράσης είναι πολύ πιο ε, προφανές και πολύ πιο ορατό σήμερα. Το κόστος ως προς τη φήμη μας για τις φρικαλαιότητες που έχουν διαπραγεί στα διάφορα μέρη. Είναι κάτι το αφόρητο και υπάρχει και κόστος που επιβαρύνει τα κράτη-μέλη σε άλλους τομείς. Το κόστος της μη δράσης εννοώ. Πρέπει να το προσεγγίζουμε το θέμα με ειλικρινή ανάλυση. Οι αποστολές για την ασφάλεια και την άμυνα ήταν ε, έμοιαζαν λίγο με τα πρώτα βήματα ενός πυγμάχου. Ε, ο προπονητής να διαλέγει κάποιους αντιπάλους για να μπορέσει ο πυγμάχος να προπονηθεί και να εξασκηθεί στο, στην αγωνιστική πυγμαχία, αλλά κρατάει μακριά πολύ ισχυρούς αντιπάλους για να μην το βγάλουν νοκάουτ. Όμως έχουμε και σενάρια υψηλού κινδύνου και θα υπάρξουν τέτοια. Θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερες απώλειες, θα μπορούσαμε να έχουμε ομήρους. Στη δεύτερη μάχη της Φαλούτζα ήταν 100 οι θάνατοι ε, μεταξύ των στρατευμάτων της Συμμαχίας. Είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε σε τέτοια κλιμάκωση αν αντιμετωπίσουμε περισσότερη αντίσταση από αυτή που περιμένει. Γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τη δράση μας, δεν θα πρέπει να παρέμβουμε εξ αρχή και να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει είναι καλύτερο. Άρα, αν ναι, θέλουμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, πρέπει να είμαστε και πιο ξεκάθαροι για τον κίνδυνο που συνεπάγεται και να έχουμε και περισσότερη διαφάνεια του τι σημαίνει αυτό από πλευράς ευρωπαϊκών απολειών ζώων ζωών, απώλειων ε, ζωών Ευρωπαίων πολιτών ή τι σημαίνει αυτό από πλευράς απώλειων ε, ε, στον τοπικό πληθυσμό, τον άμαχο πληθυσμό. Δεν θα είναι πια επιχείρηση και αποστολή τύπου Άρτεμις ή Κονκόρ, θα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Πρέπει όλα αυτά να τα ξέρουμε και να τα αποδεχθούμε. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, από τα βάθη της καρδιάς μου. Πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς. Είναι καλή συμβουλή αυτή το να ασχολείται κανείς με τον εαυτό του και να προσπαθεί να βελτιώνεται. Η μετριοπάθεια όμως δεν ταυτίζεται με την παρέτηση. Πρέπει τα λόγια μας να ταιριάζουν με τις πράξεις μας και ε, πρέπει να αποκτήσουμε τα μέσα για να πετύχουμε τις φιλοδοξίες μας. Ελπίζω σε 10 χρόνια όταν οι διάδοχοί μας θα ο οργανώσει μια αντίστοιχη συζήτηση για τα 20 χρόνια κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα, να είναι σε θέση να πούνε ότι αντλήσαν διδάγματα από τη δική μα αδυναμία, ότι στάθηκαν στο ύψο των περιστάσεων, ότι αντιμετώπισαν τι προκλήσει και ότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα θα είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο απτή και ορατή ε, τότε. Σα ευχαριστώ πολύ όλου και όλε.